μπορούμε να συνδέσουμε την παρουσία σας με την ομάδα. Σας καλωσορίζω όλους στην τελευταία σημερινή μας συνεδρίαση. Είναι εδώ και ο εισηγητής μας ο κύριος Κρόιτσμαν για να μας παρουσιάσει την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του για τα τυχερά παιχνίδια είναι η δεύτερη τέτοια έκθεση και γι' αυτό έχουμε ήδη γνώση του θέματος. Απαντάμε έτσι σε μία διαβούλευση της Κομισιόν για τα τυχερά παιχνίδια λοιπόν. Υπάρχει ο κύριος Κρόιτσμαν και οι σκιώδεις του Αμπάτ και άλλοι, δεν είναι όλοι παρόντες κύριος Φόξ όμως είναι παρόν και ο κύριος Διόν επίσης. Δίνω λοιπόν αμέσω το λόγο στον κύριο Χρόιτσμαν. Ο κύριος Φρόν από την Κομισιόν που ήταν εδώ και χθες θα μας σχολιάσει από την πλευρά της Κομισιόν. Λοιπόν, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πράσινη βίβλος, την οποία δημοσίευσε η Κομισιόν, εξετάζει πάρα πολλά ερωτήματα και τον Αύγουστο η Κομισιόν θα παρουσιάσει μία σύνοψη. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι η Κομισιόν επέλεξε μία μεγάλη βεντάλια τοποθετήσεων. Από τη μια το να μην κάνει τίποτα μέχρι την ρύθμιση. Είχαμε λοιπόν μία ακρόαση επί του θέματος και αυτή η ακρόαση κατέδειξε ότι είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν μέτρα. Γνωρίζουμε ότι, ότι ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό το επιβεβαίωσε ε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό εκφράζει και τη δική μου άποψη ότι όχι μόνο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αλλά και να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Σήμερα όλα εκείνα τα οποία αποτελούν πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να επιληθούν πάλι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σημείο υπαριθμών 1 αναφέρω ότι οι πολίτες βεβαίως και έχουν έτσι μια τάση να ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια αλλά τη μαύρη αγορά μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μεμονωμένα κρατημέλη παρότι μόνα τους προσπαθούν να καταλήξουν σε ρυθμίσεις. Την προστασία των νέων μπορεί να την επιτύχει κανείς μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε νομίζω το παράδειγμα της Φινλανδίας, της Δανίας, δεν άκουσα τη λέξη στην ακρόαση, που λένε ότι ε, σε εμά υπάρχει ένα κεντρικό σημείο καταγραφής και εκεί μπορεί κανείς να καταγραφεί μόνο αν δεν ε, προωθεί ιδιαίτερα τα, τυχερά, τα τυχερά παιχνίδια. Αυτό προστατεύει τους νέους ε, και αυτό ε, θα μπορούσε να αποτελεί και τη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, γιατί με τρόπο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ο εθισμός. Αυτά μπορεί κανενα να τα ρυθμίσει όπως σας είπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταθέτοντας μία αίτηση. Βεβαίως ε, και όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν ε, και σε ιδιωτικό επίπεδο, δεν πρέπει απαραίτητα να ρυθμίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως να λέμε μία καταγραφή, μία ταυτοποίηση και ε, αυτό σε απευθείας ε, σύνδεση μπορεί κανείς να το ε, καταπολεμήσει πάρα πολύ καλά. Είναι μια μανία, μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει και αν φτάσουμε και σε ένα σύστημα αδειοδοτήσεων πάρα πολύ καλά μπορεί να γίνει αυτό απευθείας online γιατί οι εταιρείε, τα καζίνο, οι κουλοχέρδες όπως λέμε στα ελληνικά, όλα αυτά μπορούμε να τα ρυθμίσουμε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως ε, θα πρέπει οι κανονισμοί που θα θεσπιστούν να είναι διαφανείς και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το ίδιο ισχύει και η ε, ακαιρότητα του χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων. Σήμερα το πρωί έφυξε και το θέμα του ξεπλήματος ευρώμικου χρήματος και αυτό ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί είναι σε απευθεία σύνδεση, σε ε, επίπεδο επιγραμμικό. Γι' αυτό λοιπόν για μένα το συμπέρασμα είναι ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι αποδεκτά από όλα τα κόμματα όλα αυτά μπορούν να επιληθούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πώ μπορεί να γίνει αυτό μόνο μέσω μια οδηγία. Να υπάρχει μια ελάχιστη εναρμόνιση ε, και τα κράτη-μέλη ε, να πούν ότι θέλουμε να έχουμε αυστηρότερε προδιαγραφέ. Γιατί χωρί τα κράτη-μέλη, χωρίς την επικουρικότητα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λύση. Άρα δηλαδή πρέπει να συμπεριλάβουμε στις ρυθμίσεις ε, τα κράτη-μέλη τα οποία ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να περιοριστεί η μαύρη αγορά. Και σα λέω και κάτι άλλο. Αν αν θεσπίσουμε ευρωπαϊκό κανονισμό, ε, τότε θα έχουμε εξουσία κατά της ε, μαύρης αγοράς, ε, κατά του αθέμητου ανταγωνισμού. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι σε αυτό το πρόβλημα η Ευρώπη είναι η λύση του προβλήματος και δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αρχή της επικουρικότητας. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη, αλλά είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να λύσουν μόνα τους και όλα εκείνα που μπορούν να επιληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια κατάσταση από την οποία θα υποφεληθούν όλοι. Ε, άδεια, το σύστημα της αντιοδότησης ε, θα ισχύει βέβαια για όλα τα κράτη-μέλη. Με πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο εγώ προτείνω στην έκθεσή μου είναι ότι μπορούμε να περιορίσουμε και τη γραφειοκρατία, λέγοντας ότι εφόσον υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να πούν εντάξει, δεχόμαστε τον κανονισμό αυτό, υπάρχει αυτόματη αντιοδότηση ή γίνονται οι προδιαγραφές ε, πιο αυστηρές, ε, μπορεί κανείς να πει ότι εφόσον πληρούνται και αυτές οι προδιαγραφές, αυτές ε, αποτελούν την προϋπόθεση για την απόκτηση άδεια. Ελπίζω να αποκτήσουμε ευρία πλειοψηφία και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί είμαι πεπισμένος, χωρίς ευρία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν δεν θα κάνει σχεδόν τίποτα. Η Κομισιόν τα χρειάζεται τα κράτη-μέλη. Όμως και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ακρόσης και αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, όμως λοιπόν εάν συνεργαστούν όλα τα πολιτικά κόμματα και θελήσουν να λυθεί το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν το επιτύχουμε αυτό, νομίζω θα καταλήξουμε όλοι από κοινού σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι πρόοδος ε, για ένα θέμα που όπως σας είπα μπορεί να επιληθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα εγώ ελπίζω και προσβλέπω σε ευρία πλειοψηφία. Είμαι ανοιχτό βέβαια για παρατηρήσεις ε, και προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους και ηγητέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σαφής η παρουσίαση και η ανάλυση για τη σημασία αυτής τη έκθεσης και της ενθάρρυνσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιδιώξει συνενετική λύση. Πολύ σωστή. Ο κύριος Αμπάτ. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κρότσμαν για την έκθεση που εκπώνησε και να πω ότι γενικώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο και εστερνίζομαι πολλές από τις παρατηρήσεις του και τον ευχαριστώ για την έκθεση. Για και τρία σημεία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η αγορά, η επιγραμμική online, δεν είναι όμοια με τις άλλες όπου και δεν εφαρμόζεται η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με παρόμοιο τρόπο όπω και στις άλλες αγορές. Γι' αυτό και θα πρέπει την online αγορά, την επικραμμική αγορά, να την έχουμε υπόψη με τις ιδιαίτερότητε τη. Θα πρέπει να τηρήσουμε δύο βασικές αρχές, την αρχή της επικουρικότητας. Συμφωνούμε με την ιδέα της ενεργούς επικουρικότητας. Δηλαδή να εθετήσουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά με σεβασμό της ε, εθνικής αρμοδιότητας και μια εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ώστε κάθε κράτος να μπορεί να διαφυλάξει και να διατηρήσει το κανονιστικό του πλαίσιο. Είμαι υπέρ της ενίσχυσης ε, της ε, νόμιμης προσφοράς. Μόνο έτσι, αν γίνει πιο θελκτική η νόμιμη προσφορά, θα καταπολεμήσουμε έμεσα την παράνομη προσφορά. Βέβαια, έχω εδώ μια διαφωνία. Η μείωση του γραφειοκρατικού άκθους, του διοικητικού άκθους, είναι ε, ένα πράγμα, αλλά το θέμα της ε, κοινοτικής άδειας είναι κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα και σε ό,τι αφορά τη μείωση του διοικητικού άχθους, πιστεύω και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όντω να μειώσουμε αυτό το γραφειοκρατικό διοικητικό άκτο για να ενισχύσουμε τι διασυνοριακέ συναλλαγέ. Εκτό βέβαια και αν μιλούμε για απαραίτητε διατυπώσει. Δεν μπορούμε να τι θυσιάσουμε γιατί ε, υπερασπίζουν το συμφέρον των καταναλωτών. Πάντω θέλουμε μία πλούστευση. Σε ό,τι αφορά την κοινοτική άδεια, αυτό είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας και όχι το αρχικό στάδιο. Προσοχή λοιπόν. Συμφωνούμε με την απλούστευση της χορήγησης της άδεια και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή, αλλά αυτή η απλούστευση δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει την εφαρμογή της αρχής της μη αναγνώρισης. Συμφωνώ λοιπόν με τη μείωση του γραφειοκρατικού άρθρου για να γίνει πιο ελκυστική αγορά των επιγραμμικών ε, τυχερών παιχνιδιών, αλλά να διασφαλίσουμε τα προνόμια των κρατών μελών. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα και η κατάσταση είναι περίπλοκη. Οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ ακόμη δεν επικοινωνούν μεταξύ του. Έχουμε συμβάσει εταιρική σχέση, αλλά δεν έχουμε ε, μεταξύ δύο χωρών, αλλά δεν έχουμε πραγματικά πανευρωπαϊκή συνεργασία. Αυτή τη συνεργασία και το συντονισμό θα πρέπει πρώτα να ενθαρρύνουμε μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Επίσης, ε, ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό σε σχέση με την έκθεση Σαλντεμόζε για την προστασία των καταναλωτών, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εμείνει στην ανάγκη της ακεραιότητας του αθλητισμού. Και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την αρχή και εμείς είμαστε πολύ φιλόδοξοι ως ε, συνομοθέτες και να δημιουργήσουμε το, να διοργανώσουμε το σύνδεσμο μεταξύ το, της διοργάνωσης διαφόρων αθλητικών ε, ε, οργανώσεων και της ε, προσφοράς τυχερών παιχνιδιών online ώστε να έχουμε μεν απόδοση των εργασιών, αλλά μην να είναι υπερβολικό το κέρδος και να προσέξουμε να είναι νόμιμες αυτές οι προσφορές για την ιδέα της οδηγίας. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η νομική της βάση. Αν η νομική βάση θα είναι η εσωτερική αγορά ή η προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως, κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης της οδηγίας που καταπολεμά την νομοποίηση των παράνομων ε, εσόδων, που σήμερα καλύπτει μόνο τα έσοδα των καζίνων ε, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Συμφωνώ γενικώ με τον εισηγητή. Προσοχή όμως στην ε, διαφοροποίηση μεταξύ του διοικητικού άκθους και της ευρωπαϊκής διαδικασίας χορήγησης άδεια. Και μπορούμε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι ότι φορά την ακαιρεότητα του αθλητισμού, ε, υπερασπίζοντας την αρχή του δικαιώματος ε, του στοιχήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσάς κύριε Κρόιτσμαν για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Δεν ανέμενα τίποτε λιγότερο από έναν φιλελεύθερο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση αυτή γιατί βλέπω ότι βασίζεται σε στα θεμέλια των όσων είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο το 2009. Δεν θα σας εκπλήξει όμως ότι έχω και μερικά σχόλια να κάνω. Καταρχήν, να αποσαφηνίσω κάτι. Συμφωνώ ότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στο θέμα των τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη γιατί μπορεί τα τυχερά παιχνίδια να σχετίζονται και με το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και με άλλους τέτοιους παράγοντες. Βρώμικου, βρώμικου, με συγχωρείτε. Μέχρι εκεί καλά το θέμα όμως νομίζω είναι το εξής. Με ποιο εργαλείο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις και τέτοια προβλήματα. Δεν είμαι τόσο βέβαιη ότι η λύση είναι οδηγία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συμφωνώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε πολύ καλύτερα μεταξύ χωρών μελών και γι' αυτό προτείνω να αρχίσουμε τονίζοντας ότι πρέπει η Κομισιόν να καθορίσει το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας των κρατών μελών. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει κάτι και για τους παράνομους που χορηγούν τέτοια τυχερά παιχνίδια, που λειτουργούν τέτοια τυχερά παιχνίδια. Αλλά η βασική λύση είναι τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να συνεργαστούν για να τους καταπολεμήσουν ίσως μακροπρόθεσμα να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αρκεί και ότι πρέπει να υπάρξει και κάποια οδηγία προστασίας των καταναλωτών και καταναλωτριών. Αλλά το σύστημα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αν αρχίσουμε από ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι να διευκολύνει η Κομισιόν τη συνεργασία γιατί η καταπολέμηση των παρανόμων κατα... γίνεται πολύ πιο εύκολα όταν συνεργάζονται τα κράτη. Υπάρχει το πρόβλημα του κατακαιρματισμού της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών και αυτό είναι κατανοητό εφόσον υπάρχει επικουρικότητα που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να καθορίσουν την ομοθεσία τους για τα τυχερά παιχνίδια όπως θέλουν. Έχουν, υπάρχουν διαφορετικά ήθη για τα τυχερά παιχνίδια στις διάφορες χώρες. Θα με ανησυχούσε μάλιστα αν σε αυτήν τη φάση γραφόταν οδηγία για τα τυχερά παιχνίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πολύ γρήγορα θα βλέπαμε να εφαρμόζονται ομοιόμορφοι κανόνες ενώ οι αγορές των τυχερών παιχνιδιών διαφέρουν. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για κάτι τέτοιο. Πάνω απ' όλα πάντως νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να αναγνωρίσουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μία κανονική οικονομική δραστηριότητα αλλά μία ειδική οικονομική δραστηριότητα με ιδιαιτερότητες. Και άρα πρέπει καταρχήν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών να ενισχυθεί όσοι υπάρχει και έτσι να αντιμετωπιστούν σε πρώτη τουλάχιστον φάση αυτές οι προκλήσεις. Συμφωνώ όμως ότι υπάρχει απάτη, υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ας μην τα αναφέρω τώρα όλα, συμφωνώ σε αυτά που είπατε. Ήθελα όμως να περιοριστώ στα κυριότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η έκθεσή σας είναι εξαιρετική σε πάρα πολλά σημεία της. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο επ' Όλες οι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο διαφέρουν και μεταξύ τους και εσωτερικά η κάθε μία έχουν διαφορετικές απόψεις διότι τα τυχερά παιχνίδια είναι θέμα που αφορά τα ήθη κάθε χώρας και τις συνήθειές της και άρα υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα όπως και ενδιαφέροντα και στη δική μου ομάδα το ΕΛΚ, στη δική σας δεν ξέρω. Υπάρχουν πάντως διάφορα συμφέροντα και διαφορετικά και πρέπει να πετύχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη συμφωνία και να ζητήσουμε μία προοδευτική εφαρμογή αυτών που ζητάτε κι εσείς. Τώρα μπορούν να εφαρμοστεί κάτι παραπάνω από ό,τι είχαμε πει τον περασμένο Μάρτιο. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μας που για ένα τόσο επίκαιρο και σοβαρό θέμα. Καλώ σα ευχαριστούμε για τα πολύ επικοδομητικά σχόλια που δείχνει ότι έχει νόημα να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό γιατί έχουμε σημειώσει πρόοδο σε σχέση με προηγούμενη έκθεση. Η κυρία Ρούλε, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φόξ. Μετά στην κυρία Ρούλε και μετά στον κύριο Τιόν. Έχω σημειώσει στο κατάλογο τον κύριο Βανόκ, Δεκάμπος, Μάντες, Μπουσουτήλ και Φιέλνερ Γκέπχαρτ. Άλλος κανείς, για να προγραμματίσω και το χρόνο. Ο κύριος Φόξ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την αξιόλογη έκθεσή του και την, το συνεργάσιμο πνεύμα του σε αυτό το δύσκολο ζήτημα. Φαίνεται ότι εξεπλάγει θετικά η κυρία Σάλτε από την έκβαση. Εγώ το αντίθετο, είμαι ελαφρώς απογοητευμένος γιατί περίμενα μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση του πολυφιλελεύθερου εισηγητού μας. Η κυρία Σαλτεμόζα είπε ότι ελπίζει να είμαστε πιο φιλόδοξοι ε, και να πάμε λίγο παραπάνω από το Μάρτιο του 2009. Ε, ε, εγώ θα, θα ήθελα να πιέσω τον κύριο Κρόισμαν να πάει όσο πιο μακριά γίνεται από το Μάρτιο του 2009 γιατί το σημείο φετηρίας της ομάδας μου ήταν η έκθεση της ανασχετικής μειοψηφίας ε, που γράψαμε, κύριε Πρόεδρε, και εγώ ήμουν υπέρ εκείνη τη πιο φιλελεύθερη προσέγγιση ό,τι αφορά τη ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν αρκετά τολμηρή η έκθεση αυτή και δεν καλύπτει πλήρω τι ανησυχίε του κλάδου αυτού. Γιατί εξορισμού ε, είναι διασυνοριακό ο χαρακτήρα ε, των επιγραμμικών συστηματών και παιχνιδιών και δεν υπάρχει νομική ασφάλεια αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, δεν υπάρχει αρκετή προστασία του καταναλωτή και πολλαπλασιάζονται παράνομες δραστηριότητες όπως νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε και άλλες λαθρέ και παράνομε πρακτικές. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ε, στην εσωτερική αγορά και να λάβουμε υπόψη και την προστασία του καταναλωτή. Θέλω ε, περισσότερη έμφαση σε διαδικασίες επιπαραβάσεις που έχουν ξεκινήσει κατά των κρατών μελών και που καταστρατηγούν ε, κατάφορα τις ε, διατάξεις εσωτερικής αγοράς πνίγουν την καινοτομία και εμποδίζουν τον ελεύθερο αντιγωνισμό. Και είναι κάπως ηρωνικό που ε, τα κίνητρα πολλών ε, εθνικών κυβερνήσεων για να ρυθμίσουν τυχερά παιχνίδια είναι υποτίθεται να προασπίσουν ε, τα δικά τους, τις δικές τους νομότυπες πηγές εσόδων. Αν όμως απελευθερώσουν τις αγορές, ουσιαστικά θα αυξηθούν τα έσοδά τους. Πιστεύω ότι μια σωστά ρυθμισμένη, ένα σωστό ρυθμισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το επιγραμμικό gambling, για, το, για τα online τυχερά παιχνίδια, θα έχει πολλά πλεονεκτήματα. Βέβαια, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και χέγγια και ασφαλιστικέ δικλείδε για του καταναλωτέ. Θέλουμε υπεύθυνα τυχερά παιχνίδια, προστασία των πιο ευάλωτων, δράση κατά της, ε, του ξεπλήματο ε, χρήματο και εξασφάλιση των ε, λογαριασμών online. Η κυρία Σαλντεμόζη είπε ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν είναι μια κανονική ομαλή δραστηριότητα του καταναλωτή. Αυτό είπατε κυρία Σαλτεμόζα. Α, δεν είναι, δεν είναι μια φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα, είπατε. Σας ρωτώ λοιπόν, κυρία Σχαλντεμόζε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός νεαρού ε, που αγοράζει ένα καινούριο παιχνίδι για τον υπολογιστή και ξοδεύει 40-50 ευρώ το μήνα αγοράζοντας ε, συνεχώς καινούργια παιχνίδια για τον υπολογιστή από κάποιον που λαμβάνει ε, μια συνειδητή απόφαση να, στοιχει... να ποντάρει 40-50 ευρώ το μήνα και να περνάει έτσι τον ελεύθερο του χρόνο. Μπορεί συνειδητά να επιλέξει να παίξει αυτά τα 50 ευρώ και να τα χάσει σε πόκερ που θα παίζει online ή σε άλλο τυχερό παιχνίδι μέσω του διαδικτύου. Είναι μια συνειδητή απόφαση. Ε, Μπορεί εμεί να διαφωνούμε με την επιλογή αυτή του καταναλωτή, μπορεί να διαφωνούμε ότι είναι καλό το... καλός ο τζόγος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε πρέπει να εμποδίσουμε τους καταναλωτές να το κάνουν να το επιλέξουν. Επειδή μερικοί διαφωνούν με τα τυχερά παιχνίδια, με τον τζόγο, πιστεύουν ότι θα πρέπει να εμποδίσουμε και όλο τον κόσμο να ποντάρει και να παίζει. Διαφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Και από τη στιγμή που θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη προστασία, ώστε να ε, τεθεί τέρμα στον εθισμό που δημιουργεί το τυχερό παιχνίδι. Δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε αξιολογικέ κρίσει για το πώ ε, θα επιλέγει ο κάθε καταναλωτή να εξοδέψει τα χρήματα που με τόσο κόπο έχει βγάλει από τη δουλειά του. Ευχαριστώ. I think Mrs. Felt you perhaps... Ε, κυρία Σαλντεμόζε φαίνεται πιστεύει ότι μάλλον δεν ερμηνεύτηκε σωστά. Δεν τα λέω εγώ κύριε Φόξ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι μια φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα ιδιάζοντος χαρακτήρα. Δεν ήταν δική μου ορολογία αυτή ότι δεν είναι κανονική φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα. Το ίδιο το δέκτο το είπε. Η ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι ευγνώμων για αυτά που είπε ο κύριος Φούξ, ε, γιατί πραγματικά ανοίγει το πλαίσιο και το καθορίζει μέσα αυτό που πρέπει να κινούμεθα. Ε, Βεβαίω είμαι πιο ευγνώμων στον κύριο Κρότσμαν ε, και χαίρομαι που δεν ήταν συγητής των φιλεύθερων κύριος Μάντας και που ήταν τελικά ο κύριος Κρότσμαν, γιατί θεωρώ ότι με την έκθεση τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. Χωρίς αυτή την έκθεση δεν θα το κατορθώναμε. Η βάση που καθορίζετε εσείς ανοίγει μια συζήτηση στη Γερμανία ε, που δεν θα είναι εύκολη και θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριο Φόξ ε, σχετικά με τα κέρδη και τη χρησιμότητα. Αν δείτε λιγάκι ποιος κερδίζει ε, σε ένα κράτος μέλος όπως η Γερμανία, αν δείτε ποιος κερδίζει από αυτά τα παιχνίδια, καταρχήν είναι οι ερασιτέχνες αθλητές και οι κοινοφελείς οργανισμοί. Αν αυτά ε, εισήρχονται ε, σε ένα κρατικό κορβανά με φόρο κανείς δεν θα ωφελεί το από αυτούς που ανέφερα και σίγουρα όχι οι επαγγελματικές ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Κρόιτσμαν αυτό που λέτε ε, τα έσοδα που θα πρέπει να διοχετεύονται ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη πολιτιστική διαφορά στα κράτη-μέλη. Ε, βλέπετε το πώς εννοούμε εμείς το τι πρέπει να γίνεται με αυτά τα χρήματα και πώς τα εννοούν άλλοι. Όσον αφορά τις ε, προτάσεις του κυρίου Κρόιτσμαν, ε, θίγεται την επικουρικότητα, την αμοιβαία αναγνώριση, το θέμα της προστασίας του καταναλωτή, των νέων, αναφέρεται και την ακαιρεότητα των παιχνιδιών. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί η νόμη προσφορά έναντι της παράνομης. Ε, και είμαι πρόθυμη να το πω αυτό στη Γερμανία. Αλλά για μένα τώρα τίθεται το εξή ενδιαφέρον ερώτημα. Και τελικά τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία. Αλλά διερωτώ με κατά πόσον η οδηγία είναι το σωστό εργαλείο. Καλύτερα να είχαμε ένα κανονισμό. Γιατί ο κανονισμό ε, θα ήταν πιο στοχευμένο και θα ήταν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ακριβώ μα ενδιαφέρει. Μα ενδιαφέρει, παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει και να ενισχύσει το συντονισμό των φορέων ανάμεσά τους. Επίσης, να δομηθεί καλύτερα η προστασία του καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε κατά πόσον το ενδεδειγμένο εργαλείο είναι η οδηγία ή ο κανονισμός. Πάντως και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Ε, θα πρέπει το βήμα αυτό να το ε, προστατεύσουμε σε εθνικό επίπεδο και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ε, δεν αντέχω πια όλα αυτά τα mail από τα λόμπι. Μας στέλνουν συνέχεια mail. Εγώ βέβαια έχω βρει μια στάνταρτα απάντηση που τους τη στέλνω σε όλους, ε, που τους λέω ότι έχει δηληθεί το θέμα και δεν ε, βλέπω κανένα λόγο να συναντηθώ μαζί σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως με την πρότασή σας κάνουμε το βήμα αυτό που είναι απαραίτητο που θα ε, καταστήσουν περιτές τέτοιου είδους επικοινωνίες ή έστω τουλάχιστον τα μέλη αυτά θα τα περιορίσουν κατά πολύ. Τέλος από τους κοιόντε, ο κύριος Διόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κρόιτσμαν για την έκθεση του. Θα ήθελα να επαναλάβω τη βάση στην οποία στηρίζεται η ομάδα μου, ότι δεν πρόκειται εδώ για κανονική οικονομική δραστηριότητα και ότι για μας το σημαντικό είναι να αποφεύγεται η κατάχρηση και η συνήθεια σε τέτοια παιχνίδια, ο εθισμός. Στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών η πτυχή που τονίζεται είναι η καταπολέμηση των καταχρήσεων και των εγκληματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Έπειτα ξέρουμε ότι σχετίζεται καμιά φορά η δραστηριότητα αυτή και με το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και άρα αναρωτιέμαι η ΙΜΚΟ χρειάζεται να ενισχύσει αυτή τη δουλειά της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Πρέπει να δεχτούμε πάντως ότι το οποιοδήποτε κράτος έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εφαρμόσει περιορισμούς στην, στα τυχερά παιχνίδια τουλάχιστον ηλεκτρονικά στο, από το ίντερνετ. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ένα κρατικό μονοπόλιο αν είναι προς το, για το κοινό όφελος. Δεύτερον, αφού μιλάμε για λήψη μέτρων, ανεξαρτήτως από την άποψη της Επιτροπής Δημοσιολευθεριών, εδώ το θέμα μοιάζει κάπως με τα θέματα που μας απασχολούν για την πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι εθνικά θέματα και γι' αυτό δεν θα ήθελα να υπάρξει οδηγία ούτε καν κανονισμός για θέματα που εξορισμού είναι εθνικής δικαιοδοσίας και διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, για κανονική οικονομική δραστηριότητα και άρα δεν είναι δραστηριότητα που σχετίζεται με την κανονική λειτουργία της εσωτερικής ή ενιαίας αγοράς. Δεν θα ήθελα να προσθεθεί κι άλλη νομοθεσία και να είναι γι' αυτό το θέμα. Είναι περίεργο που οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι ζητούν περισσότερη νομοθεσία. Εγώ θέλω όσο δυνατόν λιγότερη νομοθεσία και κανόνες και επιβαρύνσεις. Είμαι όμως υπέρ της συνεργασίας για την καταπολέμηση του εθισμού που μπορεί να είναι η συνήθεια στα τυχερά παιχνίδια, η καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος κτλ. Απλώς νομίζω ότι δεν εμπίπτει στην εντολή της Επιτροπής μας αλλά είναι εθνική δικαιοδοσία. Μάλιστα θα ήθελα τώρα να σας θυμίσω απλώς αγαπητοί συνάδελφοι ότι θα έρθει και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό της ε, Πολωνίας σε λίγο οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα. Έχω ακόμη 7 εγγεγραμμένους. Σας παρακαλώ λοιπόν για δύο λεπτά περίπου ο καθένας. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Απλώς για να μιλήσουν όλοι. Fiona, Mrs. Gephardt and Mrs. Kohler. Anybody else? Κανείς άλλος ή καμία άλλη. Α, ναι, τα είπαμε αυτά, από Μάντελσον και τα λοιπά. Mr. Mandelson is on here. Oh, so we'll start with Mr. Wang Lok for an indicative two minutes, Mr. Wang. Για δύο λεπτά κατά προτίμηση, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω την εργασία του κύριου Κρόιτσμαν που διαπραγματεύεται εδώ ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Η έκθεσή του ταυτίζει τους κινδύνους που υπάρχουν στη λειτουργία των τυχερών παιχνιδιών ιδίως με το ίντερνετ αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Ο εισηγητής απαριθμεί ορισμένους τομείς όπου θα μπορούσε να υπάρξει πιο αποτελεσματική νομοθεσία ή διευθέτηση. Δεν λέω ότι είναι κανονική οικονομική δραστηριότητα, αλλά σε κάθε οικονομική δραστηριότητα μπορεί να υπάρξει διευθέτηση και υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τομείς όπου χρειάζεται νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ποια είναι τα τέσσερα αυτά θέματα, οι τέσσερις αυτομείς, η καταπολέμηση παρανόμων αγορών, η πρόληψη του εθισμού, η προστασία των ανηλίκων και η διατήρηση του ήθους του αθλητισμού. Κύριε Ισηγητά, επιδείξατε μεγάλη θέληση και αποφασιστικότητα, αλλά δεν ήσασταν αρκετά φιλόδοξος. Γιατί για την πρόληψη του εθισμού, παραδείγματο χάρη, θα θέλαμε να προβλεπόταν κάτι για την, τον αυστηρό περιορισμό των διαφημίσεων, απαγόρευση χορήγησης βραβείων και επιβραβεύσεων ε, χρηματικών για τους παίκτες κλπ. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε μια απλή δεοντολογία. Φυσικά πρέπει να αφήσουμε χώρο για την επικουρικότητα, αλλά ορισμένοι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνο αν υπάρχουν κοινά και δεσμευτικά πρότυπα πανενωσιακώς όπως για την προστασία των ανηλίκων ή για την καταπολέμηση της απάτης στον αθλητισμό που είναι ποινικό θέμα. Τέλος, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα που θέτουν τα παιχνίδια στο ίντερνετ, τα κράτη-μέλη που, το που θα το ήθελαν θα έπρεπε να μπορούν να έχουν τη διάθεση να εφαρμόσουν ένα εθνικό μονοπόλιο. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να προστατεύσει καλύτερα τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντόγκ. Ήταν σαφέστατη και περιστατωμένη η παρουσίαση. Ο καθηγητής Κορέα Δεκάμπος. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Κρόιτσμαντ για την πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική και αξιόλογη έκθεση του που βάζει τις βάσεις για ένα καλό ψήφισμα. Βέβαια, έχω κάποια σχόλια και κάποιες διαφωνίες με τον εισηγητή. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να λέμε ότι υπάρχει μια δικαιολογία για την ε, εξάλληψη των κρατικών μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών. Αυτό μας λέει η ιστορία είναι ότι κάθε, χρό, κάθε χώρα έχει την ιδιαιτερότητά της. Άλλες χώρες προτίμησαν τα κρατικά μονοπόλια, άλλες όχι για τον τζόγο. Αλλά δεν νομίζω ότι μέσω του ίντερνετ θα μπορούμε να έχουμε μηχανισμό που υπεκφέγει οποιοδήποτε κρατικού ελέγχου και μπορεί να παρακάμψει όλα τα προβλήματα και όλα τα κολλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ δεν είναι το κρατικό μονοπόλιο στα τυχερά παιχνίδια. Το κεντρικό πρόβλημα που μας επιτάσσει η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι παράνομες δραστηριότητες και οι παράνομοι φορείς που χρησιμοποιούν ένα νέο τεχνολογικό μέσο για να επιτελούν τις παράνομες δραστηριότητες τους. Αυτό θα πρέπει ε, να προσέξουμε και όχι τόσο να ανοίξουμε τα κρατικά μονοπόλια ε, κανένα δεν μα εξασφαλίζει ότι δεν θα περάσουν από τα κρατικά στα ιδιωτικά μονοπόλια ή σε ιδιωτικά ολιγοπόλια. Ποιο μα εγγυάται ότι θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο, γιατί ιδιωτικά μονοπόλια ή ολιγοπόλια θα ήταν ακόμη μια χειρότερη κατάσταση, γιατί πραγματικά εκεί θα ήταν ανεξέλεγκτε ε, οι δραστηριότητε αυτών των ολιγοπόλιων. Αναφέρθηκε πολύ το ήθο και η κεραιότητα του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε αυτό το θέμα, αλλά δεν φαίνονται αρκετά αυτά τα σημεία ή δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά όσο η πολιτιστική σημασία ή ο κοινωνικός χαρακτήρας των παιχνιδιών. Γι' αυτό και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες στην έκθεση και συμφωνώ με τον κύριο Κρόιτσμαν, με τον εισηγητή που είπε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ιδέα της ενεργούς επικουρικότητας και όχι ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα, συμφωνώ με αυτό πλήρως με τον εισηγητή μας. Αλλά για ορισμένα σημεία, όπως σας είπα, διαφωνώ και θα καταθέσω τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Κορέα. Ο κύριος Μάντελς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Κρόιτσμαν για την πάρα πολύ καλή ανάλυση που παρουσίασε. Ε, σύμφωνα μαζί του σε πάρα πολλά θέματα. Ε, τα αρνητικά στοιχεία του online τζόγου ε, είναι γνωστά, τα έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή. Η Κρίστελ είχε και μια σχετική έκθεση. Ω τώρα προ τι λύσει για αυτό το πρόβλημα και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ξέπλυμα χρήματο από παράνομε εγκληματικέ δραστηριότητε. Επ' αυτού συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Κρότσμαν. Δηλαδή, ε, πρέπει να υπάρχει εθνική προσέγγιση ανάλογα με την οτροπία τη ε, κάθε χώρα. Θα ήθελα να επισημάνω λιγάκι τον τίτλο της ε, έκθεσης αυτής ε, που είναι απευθείας ε, τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση. Έτσι λέει η έκθεση. Που σημαίνει μπορεί κανείς, παραδείγματο χάρη από τον Ανδία, να χρησιμοποιήσει έναν ιστότοπο στην Κύπρο για να παίξει τυχερά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι είναι παράτοπο παράτυπο όχι βέβαια. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσον βέβαια τα χρήματα ε, θα χρησιμοποιηθούν ε, από το ε, Ολλανδικό Υπουργείου Οικονομικών ε, ή κατά πόσον τα καθούν. Έγινε λοιπόν μια σχετική ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι χάνονται περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ λόγω ακριβώς αυτών των ε, απευθείας ε, τυχερών παιχνιδιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αρνητικά φαινόμενα με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ξέπλυματος βρώμικου χρήματος. Ο κύριος Τεγιών είπε διότι χρειαζόμαστε μια εθνική προσέγγιση και αυτά που έθιξε ο κύριος Φόξ. Νομίζω εδώ πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά της οικονομικής δραστηριότητας. Ε, πράγματι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γιατί αλλιώς αφαιρούμε δικαιώματα από ε, τους πολίτες, από τους καταναλωτές. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε να λέμε ότι μία δραστηριότητα σε ένα κράτος είναι νεομιμή και σε άλλο παράνομη. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία όπως σας είπα θεωρώ ότι πρέπει να επιλύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Μπουζουτήλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ίσως να είπε ότι αυτή δεν είναι μια ε, φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα, αλλά ποτέ δεν είπε ότι οι διατάξεις συνθήκης, ε, κυρίως αυτές που αφορούν στην ελεύθερη μετακίνηση, δεν ισχύουν. Κάθε άλλο, οι διατάξεις αυτές ε, εξακολουθούν να ισχύουν. Ε, γι' αυτό λοιπόν αν δεχτούμε εξαιρέσεις για την ελεύθερη διακίνηση ε, τότε αυτές παραμείνουν εξαιρέσεις και δεν μπορούμε να ανατρέπουμε τους ε, κανόνες. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε τουλάχιστον ορισμένοι εξημών την εξαίρεση την κάνουμε κανόνα, ενώ η εξαίρεση πρέπει να παραμένει εξαίρεση. Που σημαίνει ότι οι διατάξει συνθήκε για την ελεύθερη διακίνηση εξακολουθούν να ισχύουν. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ιδιαίτερα υψηλή προστασία του καταναλωτή, που σημαίνει ότι όποιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει αυτά τα τυχερά παιχνίδια online προστατεύεται αυτό είναι η ουσία του θέματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν και διατάξεις συνθήκης. Αυτό λοιπόν ε, το επιχείρημα κατατείνει ε, στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση, το ελάχιστο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σωστό γιατί προστατεύουμε τους καταναλωτές ε, χωρίς να εμποδίζουμε την εφαρμογή των κανονισμών ε, κοινή αγοράς. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο λογικός τρόπος να προχωρήσουμε. Να λέμε απλά και μόνο ότι απαγορεύουμε αυτή τη δραστηριότητα ή βρίσκουμε προφάσεις για να την απαγορεύσουμε. Αυτό δεν λειτουργεί και δεν θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί σας λέω η εξαίρεση πρέπει να παραμένει εξαίρεση. Και τελευταίο σημείο, εμπιστοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κανονισμούς για πάρα πολλούς τομείς και οι κανονισμοί αυτοί εξαρτώνται από ένα και βασικό στοιχείο, την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εμπιστευόμαστε ένα τον άλλον ως προς την εφαρμογή των διατάξεων. Αν μία τράπεζα αποκτήσει άδεια λειτουργία σε μια α χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει και στη β. Αν ας πούμε μια εταιρεία πάρει άδεια ε, για την αεροπλοεία, τον τομέα της αεροπλοείας σε μια χώρα μπορεί να την εφαρμόσει και στην άλλη. Υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη και αφού ισχύει αυτό, γιατί να μην ισχύει και για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία ε, σύνδεση. Εκείνο που είναι διαφορετικό είναι ότι είναι διαφορετική οικονομική δραστηριότητα. Ναι, γιατί όχι. Ας προστατεύσουμε όσου καταναλωτές, όπως το κάνουμε και ε, όπως πρέπει να κάνει συμβαίνει με τα τσιγάρα. Έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες ε, ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση. για τα τσιγάρα. Απαγορεύεται η διαφήμιση, υπάρχουν πολύ αυστηρέ προδιαγραφέ για την προστασία του καταναλωτή και πολύ σωστά το κάνουμε. Όμως ε, δεν λέμε, παραδείγματος χάρη, ότι τα τσιγάρα ε, δεν, δεν επιτρέπεται να πολλούνται στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Καταρχήν είμαι Σουηδός και μέλος άλλων επιτροπών, αλλά παρακολουθώ αυτό το θέμα εδώ και μία δεκαετία. Γι' αυτό και χαίρομαι κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να το συζητάμε. Και παρακολουθώ αυτό το θέμα γιατί είδα από την πατρίδα μου τη Σουηδία ότι επικρατεί μεγάλη υποκρισία για το θέμα αυτό. Στην Σουηδία έχουμε δύο μονοπόλια, θα το ξέρετε, για το αλκοόλ, το ενόπνευμα και για τα τυχερά παιχνίδια. Και υποτίθεται ότι και τα διευθυντικά μονοπόλια υπάρχουν για να προστατεύσουν του πολίτε. Καλό αυτό. Διαπιστώνω όμω ότι το σουηδικό μονοπόλιο για τον τζόγο είναι ο πρώτο, ο καλύτερο ή ο δεύτερο ε, σημαντικό φορέας διαφημίσεων ε, στη Σουηδία. Αν τέτοιου είδους ε, διαφημίσεις θα είχαμε για το ένα, και για το ενόπνευμα, θα είχαμε διαφημιστικά σποτ του, του, του στυλ πιείτε βότκα ε, και θα γίνετε τυχεροί. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τους, ε, τον κόσμο από την εξάρτηση, γιατί νομίζω ότι οι, οι υπουργοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πιο εξαρτημένους οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από του πιο εξαρτημένου ε, στα τυχερά παιχνίδια. Και κανεί φαίνεται να μην είναι ευχαριστημένο. Ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε οι φορεί, ούτε οι πάροχοι, ούτε ε, οι καταναλωτέ. Υπάρχουν μεγάλε αβεβαιότητε και υπάρχει ασφάλεια, ε, έλλειψη ασφάλεια δικαίου, μα λένε. Ναι, αλλά έχουμε ε, νόμιμους, παράνομους παρόχους και Θεού, ε, κάποιου ε, σε γκρίζα ζώνη. Τι θα πει αυτό, ότι είναι νόμιμοι, θεωρούνται νόμιμοι σε ορισμένε χώρε και παράνομοι σε άλλε. Νομίζω ότι είτε με τι οδηγίε είτε με τις ε, προσφυγές επιπαραβάσεις, στόχο μα είναι να αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα υποβάλαμε οδηγία γιατί θα ήταν αδύνατο να συμφωνήσουν οι χώρε μέλη και το καταλαβαίνω. Αλλά τότε θα πρέπει να υιοθετήσουμε τον άλλο δρόμο. Και ελπίζω να καταλήξουμε τελικά κάπου. Δεν νομίζω ότι μία οδηγία επί επιστητού θα μας λύσει τα προβλήματα. Ας επικεντρωθούμε στα προβλήματα που μπορούμε να ε, επιλύσουμε. Και η έκθεση σωστά μιλάει για ελάχιστους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, των ιδιωτικών παρόχων, για οποιουσδήποτε. Και όποιοι έχουν άδειε να μπορούν να τις ασπίσουν και να τις ε, απολαμβάνουν διασυνοριακά. Να μην αποκλείονται δηλαδή από ορισμένε αγορές. Ακόμη και να απαγορεύσουμε τα τυχερά παιχνίδια έχει νόημα και τα μονοπόλια, αλλά όχι να γίνονται ε, κατά χρήσο σύστημα. Αν έχουμε άδειε, να μην υπάρχει επικάλυψη, να μην υπάρχει γραφειοκρατικό άκτο. Μεγαλύτερη συνεργασία χρειαζόμαστε από τι ρυθμιστικέ αρχέ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όχι να νύπτουμε τα σχήρα μα και να λέμε α κάνουν τα κράτη-μέλη ό,τι θέλουν. Θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Είστε πρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή στην Επιτροπή μας. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρχεστε ελεύθερα. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση βέβαια του τζόγου, είχαμε και μία κρόαση. Ε, υπάρχει το θέμα της ικανότητας των κρατών μελών να απαγορεύσουν το ε, online, ε, τον online τζόγο. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ε, συμμετέχει σε τέτοια online τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εφικτού στόχου και όχι να χανόμαστε σε τελείως ε, ουτοπικού. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η όλη αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έδειξε ότι η προσέγγιση του κυρίου Κρόιτσμαν είναι απόλυτα σωστή. Πολύ σωστά λέει ότι πρέπει να αφήσουμε μεγάλο περιθώριο για την επικουρικότητα γιατί οι πολιτιστικές ε, οι είναι τόσο μεγάλες ε, που δεν μπορούμε να βρούμε μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση για τα τυχερά παιχνίδια. Και αυτό πρόκειψε και από τη συζήτηση. Και θέλω να επισημάνω σε όσους ενδεχομένως το έχουν ξεχάσει ότι τα τυχερά τυχερά παιχνίδια ε, είχαν συμπεριληφθεί και στην οδηγία παροχής υπηρεσιών και εμείς ως Κοινοβούλιο είχαμε πει εξαιρούμε, αφαιρούμε μάλλον τα τυχερά παιχνίδια από αυτή την οδηγία με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται για τη μια συνήθη οικονομική δραστηριότητα, μια ιδιαίτερη για την οποία χρειαζόμαστε και ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Ε, δεν αφήνουμε τις συνήθιες ε, ρυθμίσεις της αγοράς, αλλά χρειαζόμαστε, είχαμε πει, ειδικέ απαντήσεις ε, για ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια. Εδώ πρόκειται μεταξύ άλλων για το ξέπλυμα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για το οργανωμένο έγκλημα, για την πρόληψη εξάρτησης, πρόκειται για θέματα υγείας, ε, πρόκειται για την ε, εξάρτηση ανθρώπων από άλλους ανθρώπους ε, και πρόκειται και για την διαβίωση οικογενειών όταν τα πράγματα φτάσουν σε ακραία φάση. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε κάποια λύση, γιατί δεν είναι το να λέμε το λίμα θα λυθεί ε, στο πλαίσιο της κοινή αγοράς. Κύριε Κρόσμαν, δεν ε, είμαι έτοιμη να απαντήσω κατά πόσον ε, χρειαζόμαστε οδηγία ή κανονισμό. Όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα ρυθμιστεί στο πλαίσιο είτε της οδηγίας είτε του κανονισμού. Πάντως, μετά από τη συζήτηση που είχαμε, νομίζω ότι μπορούμε να εξετάσουμε περισσότερο σε βάθος αυτά τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσω παρόλα αυτά, γιατί με πολύ μεγάλη σύνεση και προσοχή, αλλά και με ιδιαίτερη ευαισθησία, εξετάσατε το θέμα αυτό ε, και βασιστήκατε σε αυτά που είπε ο κύριος η κυρία Σαλντεμό ε, το 2009 στην έκθεσή της. Ε, άρα δηλαδή δεν χρειαζόμαστε να αρχίσουμε πάλι από το μηδέν. Υπάρχει κάποια προϊστορία και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Κόχαλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήμουν σκιώδης πριν από δύο χρόνια για παρόμοιο θέμα και ευχαριστώ τον κύριο Κρόιτσμαν για την τωρινή του εξαιρετική δουλειά. Όπως λέει και εκείνο, τα έσοδα των τυχερών παιχνιδιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πολλές φορές διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για την προώθηση της επιστήμης και της έρευνας. Και ο κύριος Φόξ αναρωτήθηκε γιατί να καταπολεμήσει κανείς τα τυχερά παιχνίδια αφού αυξάνουν τα κρατικά έσοδα. Πολλοί από εμά αναρωτιούνται γιατί, ανησυχούν γιατί το κόστος για την θεραπεία όσων είναι εθισμένοι στα τυχερά παιχνίδια ε, ίσως αντισταθμίζει, είναι ψηλότερο από το όφελος που δίνουν αυτά τα έσοδα στο κράτος. Εγώ είμαι από τη Φιλανδία κοντά στη Σουηδία και θα μπορούσα να σας πω ότι στη Φιλανδία κάνουμε πολλά σωστά πράγματα. Είμαστε σε θέση να περιορίζουμε τα τυχερά παιχνίδια τη νύχτα For the society, I και αυτά τα τέτοιου είδους μέτρα είναι πολύ σωστά γιατί δεν επιτρέπουν σε ορισμένους με πιο αδύνατο χαρακτήρα ή που έχουν αδυναμίες να εθιστούν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και πανενωσιακός. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους σας ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση, αν και υπήρξαν και ορισμένες διαφωνίες, αλλά αυτό είναι η πολιτική. Λοιπόν, ξέρω ότι σας πιέζω, αλλά ο χρόνος, ο χρόνος. Δεν μπορείτε, δεν μπορώ να πω μερικά πράγματα στους συναδέλφους. Όχι, κοιτάξτε, ναι, αλλά να μας μιλήσει και η Κομισιόν για λίγο και μετά εσείς θα καταλήξετε κανένα τέταρτο πρέπει να δώσω και στον επόμενο εισηγητή. Ο κύριος Φρόιν. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος διότι σας πιέζει ο χρόνος. Και εσείς μόνοι σας είπατε ότι Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για τα τυχερά παιχνίδια αφού ακούστηκαν πολλές, όλες οι απόψεις, όλη η γκάμα απόψεων. Η Κομισιόν χαίρεται ιδιαίτερα γιατί στην έκθεσή του κύριος Κρόιτσμαν κάλυψε όλα τα θέματα που τίθενται όπως κάναμε και εμείς κατά τη δημόσια διαβούλευσή μας. Εμείς δεν έχουμε καμία άποψη των προτέρων. Θα δούμε, θα διαπιστώσουμε πώς είναι τα πράγματα και ο κύριος Κρόιτσμαν μας είπε ότι ίσως και τον Αύγουστο να έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Αυτό είναι ίσως υπερβολικά αισιόδοξο γιατί τότε μόλις θα έρθουν οι πρώτες απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Πάντως θα δούμε τις απαντήσεις, θα λάβουμε υπόψη και τις απόψεις του Κοινοβουλίου και θα αναλύσουμε όλες τις αναλλακτικές λύσεις για να δούμε ποια είναι η καλύτερη. Το σαφές είναι και το είπαν και πολλοί βουλευτές εδώ ότι υπάρχουν πολλά θέματα επί πολλών από αυτά μπορεί να μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο και ίσως ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών των κρατών. Υπάρχει η οδηγία των υπηρεσιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά για καλύτερη συνεργασία, διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών και για τα τυχερά παιχνίδια. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Για να δούμε και εμείς αν χρειάζεται νομοθεσία ή όχι. Πάντως η Επιτροπή είναι ανοιχτή, αναμένουμε τη, με το αποτέλεσμα της μελέτης στην πράσινη βούλο τη δική σας έκθεση και θα δούμε. Δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο, τοποθετηθώ αυτά που άκουσα. Με τον κύριο Άλμπερτ ξεκινάω. Ε, η αμοιβαία αναγνώριση είναι θέμα αδειοδότησης ε, πολλοί παραπονέθηκαν ότι δεν είχα πολλές φιλοδοξίες, θα μπορούσα να προχωρήσω περισσότερο, θα το έκανα, αλλά υπάρχει αρχή της επικουρικότητας και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Αυτή είναι η βάση και η δική μου προσπάθεια είναι να ε, μην βασιζόμαστε στην προαιρετική συνεργασία. Αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί βεβαίω ε, οι Μαλτέζοι ενδιαφέρονται να εισπράττουν ε, χρήματα και οι Γερμανοί επιθυμούν να εισπράττουν και εκείνη τα χρήματα που δαπανώνται στη Μάλτα. Κυρία Ρουλέ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανονισμό ή όχι, ό,τι θέλετε. Είμαι ανοιχτό. Και όλα αυτά που είπατε ας τα λύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, αυτό που κάνουν οι Φινλανδοί, ότι δεν πρέπει κανείς ε, να προσελκύεται ε, με χρήματα ή οτιδήποτε άλλο και αυτό ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει την εξάρτηση από το τζόγο και αυτό ε, μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό τα έφυξα όλα αυτά στην έκθεσή μου. Όλα αυτά τα οποία επιθυμείτε διακαώς και εσείς και οι σοσιαλδημοκράτες όλα αυτά να ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι θα κάνουμε ένα βήμα περισσότερο. Και έτσι θα μπορέσουμε μπορέσουμε να σπάσουμε και τα μονοπόλια. Όμως ε, τα κράτη-μέλη, όπως σας είπα, είναι κίνα που ε, ε, δεν μπορούν να λένε ότι ας πούμε κάποιος αποκτάει άδεια μόνο στη Μάλτα και όχι στη Γερμανία αν η αδειοδότηση ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντάξει αυτά που ισχύουν για τη Μάλτα να ισχύουν και την Αγγλία οι Γερμανοί αν λένε ότι θέλουμε υψηλότερες προδιαγραφές ε, τότε και αυτό να λαμβάνεται υπόψη στην αδειοδότηση και στη γραφειοκρατία ε, να πούμε ότι πράγματι πρέπει να καταπολεμηθεί όμως δεν θα υπάρχουν αυτόματες αδειοδοτήσεις ε, γιατί τότε θα αποτύγχανε η αρχή της επικουρικότητας. Και αυτό που είπε και ο συνάδελφος ε, με τους ε, φορείς οργάνωση αγώνων. Αυτοί θα αποφασίζουν μόνοι τους κατά πόσο θα τα διοχετεύουν τα χρήματα στον αθλητισμό ή στην εκτροφή αλόγων ή θα βάζουν τα χρήματα στα ταμεία τους. Είναι δική τους απόφαση και δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε τίποτα ούτε με οδηγία ούτε με οτιδήποτε άλλο. Να μην λέμε πράγματα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, να λέμε αυτά που είναι εφικτά. Και όπω σα είπα και η ε, κυρία Σάλντε Μόζα, ε, σκεφτείτε τα αυτά που επιθυμείτε ε, ε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, σύγχρονα προγράμματα ή όχι. Εγώ το σκέφτηκα. Μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να προχωρήσουμε. Να κερδίσουν όλοι δεν γίνεται γιατί οι Μαλτέζοι ε, θα ήθελαν να κρατήσουν τις, ε, τους φορείς ε, τυχερών παιχνιδιών στην πατρίδα τους και οι Γερμανοί θέλουν να κρατήσουν τα λεφτά στη δική τους την πατρίδα. Ε, ας πούμε ένα άλλο θέμα οι Ασιάτες που έρχονται εδώ και μας κατακλείζουν με παράνομες διαδικασίες αυτούς πώς θα τους αντιμετωπίσουμε και πάλι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά κύριε Ντεγιόγκ την εξάρτηση από τον τζόγο και αυτό μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει γιατί ε, το να καταγραφεί κανείς και να αναγνωριστεί σε 27 διαφορετικές χώρες αυτό δεν σημαίνει καταπολόμηση μόνο αν υπάρχει ε, κεντρική καταγραφή και όταν υπάρχει η ε, επιγραμμική διασύνδεση και καταγραφή, τότε θα ξέρει κανείς ε, και ποιο ε, παίζει τυχερά παιχνίδια και ποιο όχι. Όχι να παίζουν τυχερά παιχνίδια αυτοί που παίρνουν το επίδομα ανεργία στη Γερμανία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει πράγματι να προχωρήσουμε αυτό που έχει σημασία είναι να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Ε, πλέον τα πράγματα έχουν σημειώσει πρόοδο, να πει ο καθένα ε, τι επιθυμεί και μετά θα συζητήσουμε να δούμε κατά πόσο είναι καλύτερα να υπάρχει οδηγία ή κανονισμό. Αλλά ο στόχο είναι ότι μπορεί να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ρυθμίζεται και μετά από αυτό να ισχύει η αρχή τη επικουρικότητα. Κύριε Κρόιτσμαν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που προκαλέσατε έτσι μια ε, πολύ ζωντανή συζήτηση. Είναι ίσως ε, η πιο ενδιαφέρουσα που είχαμε εδώ και αρκετό καιρό γιατί είχαμε και πάρα πολλούς ε, παρόντες. Και νομίζω ότι εσείς είσαστε ο κατάλληλος ε, για να ε, προκαλέσετε όλη αυτή τη ζωντάνια και να ε, φέρετε και εδώ τόσους πολλούς συναδέλφους. Ελπίζω η Κομισιόν να επιληφθεί του θέματος. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Και τώρα, καθαρά τυπικά η διορία είναι 18 Ιουλίου για Τάθεση τροπολογίων θα ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου. Και στην περίπτωση που θεωρείται ότι είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα είναι διότι θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δική μας την άποψη όταν θα δώσει την απάντηση της μέσω της πράσινης βίβλου. Ε, τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό που δεν είχαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή ε, για τον κύριο Έρια Σεβαρία που ζήτησε να προεδρεύσει ε, τις ομάδες Εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μας ε, παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ πρωτοπόρα πρωτοβουλία της Επιτροπής. Είναι μια πρωτοβουλία που αφορά όλες ε, τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Σεβερίας να προεδρεύσει σε αυτήν την ομάδα εργασίας και αυτό που θα κάνουμε είναι να προσφέρουμε τη δυνατότητα για συζήτηση μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Όσον αφορά τώρα στην Επιτροπή, βλέπω ότι η κυρία Λαμότ ε, από την ε, πολιτική για online συνδέσεις είναι εδώ, αλλά εσείς ε, ο επόμενος ο συνάδελφός της που ήταν ε, αρμόδιος για τα τυχερά παιχνίδια τώρα έχει μετατεθεί και, και πάλι σας ε, καλωσορίζουμε με τη νέα σας αυτή ιδιότητα. Ο κύριος Σεβερία θα μας κάνει μια παρουσίαση θα ήθελα να επισημάνω στους συναδέλφους ότι είναι μια έκθεση από το παλιό κόμμα ε, γι' αυτό λοιπόν ε, ε, για το θέμα του λογότυπου, αυτό θα το δούμε λιγάκι για τις μελλοντικές παρουσιάσεις, ίσως για το μέλλον να αναθέσουμε σε κάποιους να βρουν ένα νέο λογότυπο. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Σεβερία, έχετε το λόγο για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ. Μια και αναφερθήκατε στο λογότυπο, να σας πω γιατί αναφέρετε το λογότυπο του ΕΛΚ. Ε, η παρουσίασή μου είναι η προσωπική παρουσίαση, δεν είναι το έγγραφο των συμπερασμάτων και είναι κάτι που απαιτείται διαδικαστικά από το κόμμα. Θα ήθελα να, να σας ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση για το ενδιαφέρον που δείξετε για αυτή την έκθεση που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας που συστήσαμε το προηγούμενο Φεβρουάριο. Πέντε μήνες μετά η παγκόσμια κρίση έχει επιδεινωθεί και η κατάσταση σε ορισμένες χώρες μέλη είναι πολύ ανησυχητική. Μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει μία και μόνο Ευρώπη, μία ή μία Ευρώπη απέναντι στην κρίση. Η κρίση ε, δείχνει πόσο διαφορετικά είναι τα συμφέροντα των κρατών μελών και το θέμα είναι να βρούμε ποιες ε, κοινέ ευθύνες θα αναλάβουμε και ποια όρια θα θεσπίσουμε. Είμαι πεπισμένος ότι η έξοδος από την κρίση βρίσκεται στον ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό και έχει νόημα να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε μια πραγματικά ε, ψηφιακή εσωτερική αγορά. Όπως ξέρετε, ήδη το Φεβράριο είδαμε στην Επιτροπή αυτό το σενάριο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν είναι και πολύ ε, ενθαρρυντική. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και τεχνικά και εμπορικά κολλήματα, μια παροχημένη νομοθεσία που δεν δίνει ενάβσματα ούτε στους ε, επιχειρηματίες ούτε στους ε, ελεκτικούς φορείς. Και υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη ενημερότητας, κάτι που δημιουργεί μια δυσπιστία και ανασφάλεια στο καταναλωτή. Αυτή η εικόνα δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματικά δεν μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως ε, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μια κανονιστική ε, διευκρίνηση και κάποιες ε, ελεκτικές υπηρεσίες που θα δίνουν εχέγγυα για τους αγοραστές, για τους καταναλωτές, λογιστικούς κανόνες διαφανής και υπέρβαση των τεχνικών φραγμών με διασυνδέσεις ε, ε, μεγάλης ε, ταχύτητας. Έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες και καταναλωτές. Για να υλοποιηθεί όμως αυτή η εσωτερική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να κάνουμε έναν προσδιορισμό των προσεγγίσεών μας και να βρούμε κάποιες διεξόδους στα προβλήματά μας. Νομίζω ότι ο πιο γρήγορος δρόμος είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα που θα είναι ένα εγγυημένο εμπορικό σήμα που θα εξασφαλίσει διαφάνεια, σαφήνεια και νομική ασφάλεια για τους καταναλωτές στις διασυνοριακές συναλλαγές υπό το σήμα ΕΕΟΥ, ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα έχουμε πραγματικά μια λογοδοσία. Θα ενημερώνεται ο χρήστης λεπτομεριακά για όλα τα θέματα που αφορούν την συναλλαγή που θέλει να πραγματοποιήσει, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ομάδα εργασίας που σύστησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς συγκέντρωσε και εκπροσώπους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής και εκπροσώπους των ε, ο ε, καταναλωτών αλλά και εμπειρογνώμονες ηλεκτρονικού εμπορίου. Και τα συμπεράσματα που σας παρουσιάζουμε καλύπτουν 7 σημεία που θα ήθελα να σας απαριθμίσω. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προστασία των δεδομένων, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ΦΠΑ, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ενίσχυση των δικαιωμάτων και τέλος το ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα. Ας ε, αναλύσουμε διεξοδικά καθένα από τα σημεία αυτά. Όπως βλέπετε στην παρουσίαση, έχουμε για καθένα από τα σημεία αυτά μια επισκόπηση της κατάστασης και τις προτάσεις της ομάδας εργασίας. Νομίζουμε ότι αυτός είναι καλός τρόπος για να δούμε πού βρισκόμαστε και να δείξουμε το δρόμο που θέλουμε να διανύσουμε. Εγώ θα περιοριστώ στην απαρίθμηση των συμπερασμάτων, γιατί δεδομένη της κατάστασης ε, ε, θα πρέπει σε αυτά να επικεντρωθούμε. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταρχήν η έγκριση οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών συνιστά πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη ασφάλεια δικαίου για πολλά ζητήματα. Χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα εναλλακτική επίλυση των επιγραμμικών διαφορών. Επίση, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα των Δικαιωμάτων online, Όπω αναφέρεται στο ψηφιακό πρόγραμμα για την Ευρώπη, καθώ και ένα δεντολογικό κώδικα για του χρήστε των επιγραμμικών υπηρεσιών. Ε, πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε ενάυσματα και πόρους στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών. Να δώσουμε έμφαση στην δημιουργία συγκριτικών ιστοτόπων, προϊόντων με πολυγλωσσικά συστήματα για να είναι εύχριστα τα συστήματα αυτά για να κάνουν το σύγκριση των τιμών οι Ευρωπαίοι. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ένα χαμηλό ποσοστό μας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν ε, ιστοσελίδα ή πολλούν τα προϊόντα τους ε, μέσω του διαδικτύου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να γίνει ο πυρήνα των δραστηριοτήτων του, παρέχοντά του ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και καλύτερη πρόσβαση στου πελάτε. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε στη διάθεσή του κάποια εργαλεία που να διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα, το δίκτυο στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το πρόγραμμα για, την, για τις, ψηφιακές δεξιότητες, ο ξεχωρισμός των μηχανισμών online δημόσιων συμβάσεων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και επιπλέον να ενημερώσουμε καλύτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ευνοήσουμε τη συμπερίληψή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω ενημερωτικών εκστρατιών. Η ιδιωτική σφαίρα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημα των καταναλωτών κατά τη στιγμή της, των αγοραπολισιών online και αυτό σίγουρα αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η κοινοτική νομοθεσία είναι άνηση. Η ομάδα εργασία υποβάλλει τέσσερι προτάσει για την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε καταρχήν μια εναρμόνιση και εξυγχρονισμό των κανόνων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο προβλέψιμο νομικό περιβάλλον και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που ισχύουν για τα δεδομένα. Διαφάνεια των δεδομένων για το πώς ε, γίνεται συγκέντρωση και φύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, εξασφάλιση διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων ανα πάσα στιγμή. Επίσης, να προβλεφθεί η διαγραφη δεδομενων να πασα ενημέρωση καταγγελίας των παραβιάσεων. Θα πρέπει να μειώσουμε και το διοικητικό φόρτο και να πλουστεύσουμε τις απαιτήσει κοινοποίηση, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Τέλος, σημαντικό είναι να προσαρμόσουμε την ομοθεσία για την προστασία δεδομένων στις νέες μελλοντικέ προκλήσεις και καινοτομίε, όπως ε, το cloud computing, όπου μέσω το ίντερνετ και εξωτερικών υπηρεσιών συγκεντρώνονται πληροφορίες και γίνεται διανομή προγραμμάτων, πόρων κτλ. Η ομαλή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τι πωλήσει εξ αποστάσεω. Διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου διατίθενται μόνο μέσω του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Μπορούν να αγοραστούν μόνο στο εξωτερικό και μάλιστα μερικέ φορέ σε χαμηλότερε τιμέ. Παρ' όλα αυτά και οι πολιτέ και οι καταναλωτέ θεωρούν τη φυσική παράδοση των προϊόντων αυτών ω φραγμό. στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο η παράδοση δεμάτων από μία χώρα σε άλλη ε, Προποθέτει πολύ υψηλότερα τέλη από ό,τι γίνεται η παράδοση στο εσωτερικό μια χώρα και αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλού και διάφορου λόγου. Προτάθηκαν πολλέ και διάφορε λύσει από την άποψη αυτή στην ομάδα εργασία. Για παράδειγμα, ομοιόμορφου και απλού κανόνε για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε στο διασυναριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίω ε, των κανόνων για το ΦΠΑ. Αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με τι υπηρεσίε αποθήκευση. Ποιες ε, είναι οι εφαρμοστές νομοθεσίες, ε, ποιοι νόμοι και ποιες χώρες χείουν, ποιες χώρες ο ΦΠΑ εφαρμόζεται. Επίσης, ομοιόμορφη οικολογική φόρη και τέλη χρήση οδικού δικτύου, όπως το σήμα τελών κυκλοφορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωβινιέτ. Ε, γιατί έτσι ίσως αυξάνονται οι χρεώσεις και το κόστος για τους πελάτες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Διευκρίνηση των δικαιωμάτων αποστολή και βελτίωση των εξή στοιχείων. Αξιοπιστία, ταχύτητα τη αποστολή, φιλική εξυπηρέτηση του πελάτη και καλή πολιτική επιστροφών. Ω προ το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ ίσω είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, έχουμε και το πιο περίπλοκο εμπόδιο σε ό,τι αφορά την αναζήτηση κάποιων κοινών στοιχείων. Αν δεν καταλήξουμε όμως σε συμφωνία για τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή του ΦΠΑ, τι εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν, ίσως πανευρωπαϊκή εμπορικός φόρος, ε, ίσως υπό το σήμα, το εμπορικό σήμα, που θα χρηματοδοτήσει τα κοινωτικά θεσμικά όργανα. Αυτό ίσως είναι μια εναλλακτική λύση που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι διάφορες προτάσεις που συζητήθηκαν στην ομάδα εργασίας είναι εξή. Απλούστεροι και ομοιόμορφοι κανόνες για τον ΦΠΑ επί των εξαποστάσεων πωλήσεων. Μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύσταση μόνο απευθυντικής θηρίδας, one stop shop, μια πρόταση που έγινε το 2004. Αποσαφήνιση της δικαιοδοσίας που ισχύει για ζητήματα ΦΠΑ σε σχέση με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και διερεύνηση των δυνατοτήτων μείωση του ΦΠΑ ή απαλλαγής από το ΦΠΑ στις διασυνοριακές online συναλλαγές προστασία δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία ε, και καταπολέμηση τη απομίμηση, παραποίηση και πειρατεία. Σημαντικέ προκλήσει και επίση πολύ σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα εξασφαλίζει ένα νομικό πλαίσιο που θα βελτιώνει και θα επικαιροποιεί την ε, νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση και εκτέλεση των πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να προσαρμοστούμε την ε, ψηφιακή οικονομία του 21ου αιώνα. Ποιε είναι οι προτάσει τη ομάδα. Αναθεώρηση τη οδηγία σχετικά με την επιβολή του, του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία που αναμένεται το 2012 για τη βελτίωση τη επιβολή και την προσαρμογή τη στην ψηφιακή εποχή. Αναβάθμιση του νομικού πλαισίου εντό του οποίου λειτουργούν τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Πρόταση και εφαρμογή αποτελεσματική νομοθεσία για την απλούστευση τη συλλογική διαχείριση στην Ευρώπη και έναρξη διαλόγου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ε, online διάδοσης οπτικοακουστικών έργων. Τέλος, το ενιαίο σήμα, ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνη. Η ομάδα ε, συστήνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων για να διαμορφώσουν ε, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του σήματος εμπιστοσύνης και η εκπόνηση ενός δεντολογικού κώδικα για να δημιουργηθεί ένα σήμα εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο που θα είναι σημαντικό ώστε αυτή, αυτό το σήμα εγγύησης να είναι ορατό, ε, αποτελεσματικό και διαφανές και κάτι τέτοιο προϋποθέτει φυσικά έναν προϋπολογισμό ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματικό αυτό το σήμα. Πιστεύω ότι το ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα θα πρέπει να, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποτελέσει ένα νομοθετικό όχημα που θα περιλαμβάνει τις οδηγίες ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενημερώνοντας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο τους εμπόρους όσο και τους καταναλωτές. Και θα πρέπει ταυτόχρονα να μας επιτρέψει ε, προσαρμογή στις ραγδαίες εξελίξεις της κοινωνίας, γιατί πραγματικά η τεχνολογία προχωρεί με ηλικιώδεις ρυθμούς και δεν θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να μένει πίσω. Στον ε, ε, ηλικιώδη ψηφιακό κόσμο ε, του 21ου αιώνα θα ήταν τρέλα κάθε φορά που γίνεται μια σημαντική αλλαγή να προτείνουμε συνέχεια μεταρρυθμίσεις. Γιατί τις μεταρρυθμίσεις θα μας κάνουν να χάσουμε το χρόνο και την ενέργειά μας και πολύ γρήγορα θα χάνουν την επικαιρότητά τους, γιατί θα πρέπει με τους νέους καιρούς να σταματήσουμε την, ε, την κανονιστική ανελαστικότητα και να βρούμε πιο ευέλικτες ρυθμιστικές λύσεις. Και για να υλοποιήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη, στην ομάδα εργασία ε, εντοπίσαμε κάποια θέματα που χρήζουν ιδιαίτερη παρακολούθηση. Καταρχήν, πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού της ενιαίας αγοράς, των διαφορών του ΦΠΑ και την έλλειψη εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών και των πελατών. Επίσης, θεωρούμε θεμελιώδους σημασία να συνδέσουμε την ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου με την πράξη της ενιαίας αγοράς. Και φυσικά και γιατί όχι, να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και να ξεκινήσουμε την συζήτηση ενός ειδικού καθεστώτος για ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε το ηλεκτρονικό εμπόριο να γίνει σαν ένα νέο κράτος μέλος, το ευρωπαϊκό, ένα ψηφιακό κράτος μέλος, για να ξεπεράσουμε επιτέλους ε, τους ισχύοντες φραγμούς. Τέλος, ήθελα να σας εκφράσω τη βούληση και την επιθυμία της ομάδας εργασίας που σας υπέβαλε τα συμπεράσματα που σας παρουσίασα σήμερα, να συνεχίσουμε με τη βάση αυτή και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα για να προχωρήσουμε γρήγορα και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα επίσημα να σας ζητήσω εδώ σήμερα να συνεχίσετε την εντολή της ομάδας εργασίας της ΣΥΜΚΟ για το ηλεκτρονικό εμπόριο για να συζητηθούν συνεχιστούν οι συζητήσεις και να περιληφθούν και άλλα θέματα που χρήζουν εξέτασης και που εξαιτία της έλλειψης χρόνου δεν μπορέσαμε να περιλάβουμε στις τέσσερις αυτές συνεδριάσεις. Θα ήθελα επίσημα να ζητήσω τη συνέχιση της εντολής αυτής της ομάδας εργασίας και η έγκρισή τη να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη τη επόμενη συνεδρίασης των συντονιστών της Επιτροπής Εσωτερική Αγορά και προστασία του Καταναλωτή. Και επαναρχόμαστε στην αρχή, γιατί τα συμπεράσματα αυτά είναι μία απλή πρόταση βελτίωση τη κατάσταση που ουσιαστικά ζητεί συνέχιση τη εργασία για να υπερβούμε του υπάρχοντε φραγμού. Γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και βασικό έργο των θεσμικών οργάνων είναι να υπερκεράσουν αυτά τα εμπόδια και του φραγμού για να επιτρέψουν μία ε, πραγματική ενοποίηση του εσωτερικού ψηφιακού εμπορίου. Μόνο έτσι θα προωθήσουμε την κατανάλωση στην Ευρώπη. Με ένα λειτουργικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει ενωμένοι να διαμορφώσουμε ένα όχημα που θα είναι ανθεκτικό στις, στις ε, κανονιστικές αλλαγές. Θέλουμε ένα όχημα που θα είναι αντίδοτο και θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατά τη γνώμη μου το όχημα αυτό είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα του πανευρωπαϊκού ψηφιακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτή είναι η διέξοδος από την κρίση και έχει ψηφιακή μορφή. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Άριας και σας και όλα τα μέλη της ομάδας σας για την τεκμηρίωση που μας δώσατε. Στην πρώτη συνεδρία των συντονιστών μας, μετά τις διακοπές, θα δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα χειριστούμε την πρότασή σας. Ήδη έδωσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Πολωνίας ένα αντίγραφο που δείχνει ότι συνδέουμε το δικό σας θέμα με τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα και στο προσεχές βήμα που θα οργανωθεί η συζήτηση για την εσωτερική αγορά θα το λάβουμε ιδιαίτερο υπόψη. Τώρα είναι ιδιαίτερη χαρά μου κυρίες και κύριοι που καλωσορίζω εδώ επισήμως για πρώτη φορά ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Δέμαρ Παύλακ που θα προεδρεύσει και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητος ως Υπουργός Οικονομικών. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα μετά την Ουγγρική Προεδρία που βλέπουμε ότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ξαναοργανώνεται. Επίσης καλωσορίζω την κυρία Μαλγκορζάτα Κρασνοντέμψκα Τόμκελ που είναι πρόεδρος του γραφείου ανταγωνισμού και καταναλωτών. Όσοι πήγατε μαζί μας στην επίσκεψή μας στη Βαρσοβία, μπορεί να θυμάστε ότι την είχαμε συναντήσει και τότε και είχαμε συζητήσει θέματα προστασίας καταναλωτών και καταναλωτριών καθώς και θέματα επιτήρησης των αγορών εποπτείας των αγορών και είναι και ο κύριος Μάρσιν Κόρελετς εδώ που είχε συμμετάσχει στην πρώτη συζήτησή μας, διάσκεψή μας για την ενιαία αγορά και ελπίζουμε να συμμετάσχει και στην επόμενη 2 με 4 Οκτωβρίου. Θα συνεργαστούμε φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερο με την Προεδρία Ξέρουμε ότι την ενιαία αγορά και την προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών θα τις έχετε από τις κύριες προτεραιότητές σας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σας δίνω το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Οι συνάδελφοι σίγουρα θα θελήσουν να σας θέσουν και ερωτήματα. Πρώτα οι συντονιστές και συντονίστριες και μετά τα υπόλοιπα μέλη. Ορίστε κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή γιατί εκ μέρους της Πολωνικής Προεδρίας ε, θα σας παρουσιάσω τα σχέδια και τις προθέσεις της Πολωνικής Προεδρίας ε, σε ό,τι αφορά τους τομείς αρμοδιοτήτων και ενδιαφερόντων της Επιτροπής ε, Εσωτερικών Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή το θέμα τη προστασία του καταναλωτή, τη θέση της πολωνικής κυβέρνησης παρουσιάσει η κυρία Κρασνοντέμσκα Τόμκιελ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δέκα θέματα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικά για την Πολωνική Προεδρία. Το πρώτο είναι η πράξη της ενιαίας αγοράς, κατόπιν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το τρίτο θέμα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Το τέταρτο η οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Το πέμπτο είναι η πρόταση για, την, για τον κανονισμό ευρωπαϊκής τυποποίησης, το θέμα του κανονισμού για, του, για τα οχήματα με κινητήρα, το έβδομο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την εισαγωγή προϊόντων στην εσωτερική αγορά και την προσαρμογή 10 οδηγιών. Το 8ο είναι η πρόταση για τον κανονισμό περιαγωγής και το θέμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις συμβάσεις παραχώρησης και τις δημόσιες προμήθειες. Ενώ ε, δέκατο θέμα είναι ο κανονισμό για την εκτέλεση από τι θελωνιακέ αρχέ των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα στο πρόγραμμα τη Πολωνική Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τα γενικά ζητήματα, η Πολωνική Προεδρία επικεντρώνεται σε τρία σε τρεις κυρίως άξονες και κατευθύνσεις, την ε, ολοκλήρωση στην Ευρώπη, την ε, ασφάλεια στην Ευρώπη και μια ανοιχτή Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την όλο και πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη, η ολοκλήρωση είναι σημαντικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης. Ασφαλέστερη Ευρώπη. Όταν μιλάμε για ασφαλέστερη Ευρώπη, εννοούμε την ασφάλεια τροφίμων, την ασφάλεια της ενέργειας και την άμυνα. Και το τρίτο, ο τρίτος άξονας, η τρίτη κατεύθυνση είναι μια Ευρώπη όλο και πιο ανοιχτή, δηλαδή με το βλέμμα στραμμένο προς τις νέες χώρες που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, για παράδειγμα, θα υπογράψουμε τη Σύμβαση Ένταξης τη Κροατία, που τον Ιούνιο στη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας ολοκλήρωσε τις προεδοξιακέ διαπραγματεύσεις και έκλεισε τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων και η Κροατία θα είναι το επόμενο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα για την Πολωνία είναι πολύ ευχάριστη αυτή τη στιγμή γιατί λένε ότι τον 7ο αιώνα οι Κροάτες μετακόμισαν στην Κροατία, με, με, στην, στο Λβόβ της Ουκρανίας, της σημερινής Ουκρανίας και εδώ και πολλά χρόνια οι Σλοβαίνοι και οι Κροάτες τουρίστες ε, περιφέρονται σε αυτή την κοινή Ευρώπη. Οπότε είναι επιστροφή ουσιαστικά στην κοινή Ευρώπη και κάτι τέτοιο θα μας ε, ανοίξει τις εμπορικές μας σχέσεις και συμφωνίες ε, γιατί οι εμπορικές συμφωνίες είναι σημαντικές ε, και για τους γείτονες αλλά και με τους υπόλοιπους εταίρους παγκοσμίως. Επανέρχομαι τώρα στα θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο την Επιτροπή σας, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Πολωνία είναι γνωστό ότι είναι ε, μεγάλος υπέρμαχος της εσωτερικής αγοράς και στην εσωτερική αγορά θεωρούμε ότι υπάρχει η, δυνατότητα ανάκαμψης από την κρίση και προώθησης της αηφόρου ε, οικονομικής ανάπτυξης. Και μάλιστα θα είμαστε ο πρέσβης ε, του, της εσωτερικής αγοράς, της ιδέας της εσωτερικής αγοράς και αυτό το ρόλο θα παίξουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και σίγουρα η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς αποτελέσει προτεραιότητα Τη Πολωνική προεδρία, γιατί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μοχλό ανάπτυξη κατά τη γνώμη μα. Θα περάσω τώρα στα επιμέρου θέματα. Το πρώτο, όπω σα είπα, ήταν, είναι η πράξη τη ενιαίας αγορά. Πρόκειται για ένα εμβληματικό σχέδιο τη εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι και στη διάρκεια τη ε, Ουγγρικής Προεδρία, αλλά και στην προηγούμενη Βελική Προεδρία, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα υιοθέτησε συμπεράσματα με βάση το έγγραφο αυτό, επιβεβαιώνοντα ε, την ε, δέσμευσή τους ε, για να δώσουν νέα όθηση στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αλλά και η Πολωνική Προεδρία θεωρεί το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και στόχος μας είναι να εγκαινιάσουμε στο Συμβούλιο ε, τις συζητήσεις για αυτούς τους 12 μοχλούς της εσωτερικής αγοράς ώστε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στις εργασίες, ε, προετοιμάζοντας το, το, τις νομοθετικές πράξεις που κατά πάσα πιθανότητα θα υποβληθούν στη διάρκεια της Θενέζικης και της Κυπριακής Προεδρίας. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τις δικές σας εμπειρίες και γνώσεις και στα πλαίσια της συναπόφασης θα έχουμε στενή συνεργασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ θερμά την κυρία Σάντρα Καλνιέτε τον κύριο Αντώνιο Φερνάντο Κορέα Δεκάμπος και τον κύριο Κρίστιαν Σίλβα Μπουσόη για την εκπόνηση εκθέσεων σε ό,τι αφορά τρεις πυλώνες της πράξης ενιαίας αγοράς. Αυτές οι εκθέσεις που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλλουν τα μάλα στη συζήτηση για το μέλλον της εσωτερικής αγοράς και μάλιστα οι συστάσεις σας ε, αντικατοπτρίστηκαν και στην τελευταία έκδοση της ανακοίνωσης. Δεύτερος σημαντικός τομέας είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και μάλιστα ακούσαμε ένα απόσπασμα της συζήτησης ή της παρουσίασης που έγινε για το θέμα αυτό που είναι σημαντικό και για την Πολωνική Προεδρία γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση και αξιοποίηση των ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες και να άρουμε τα νομικά και διοικητικά εμπόρια, να ενισχύσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης των χρηστών και την εμπιστοσύνη τους ε, στην πραγματοποίηση τέτοιων συναλλαγών. Και εδώ προσβλέπουμε στη συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Επιτροπής ΙΜΚΟ για τα θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου υπό την Προεδρία του κυρίου Ετσεβαρία ο οποίο πριν από λίγο σα παρουσίασε τα συμπεράσματα αυτή της ομάδας εργασίας ε, και την έκθεση τη ομάδα εργασία. Μα ενδιαφέρει πολύ και η δέσμευση για το θέμα αυτό και μα ενδιαφέρουν και οι συστάσει σα. Θα ήθελα εδώ να ε, αποτίσω φόρο τιμή στην Ουγγρική Προεδρία που συνέβαλε στη διεκπαιρέωση των δραστηριοτήτων της οδηγίας, των διαπραγματεύσεων της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή γιατί πραγματικά έτσι τίθενται τα θεμέλια για τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές ε, και θα βοηθεί έτσι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγώ, εκτός πολιτικής, εργάστηκα σε μια επιχείρηση που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχω και τέτοια εμπειρία. Δεν θα πρέπει να μελούμε λοιπόν τις σχέσεις με τους ανθρώπους, τις κοινωνικές σχέσεις. Και όταν θέλουμε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι μερικές φορές στερούμε από τους ε, μεσάζοντες, τους broker, ε, την ευκαιρία δραστηριοποίηση. Γιατί είναι πλατφόρμα επικοινωνίας, αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι που εξασφαλίζουν ε, άμεσες επαφές με τους πελάτες, με τους καταναλωτές και η συμμετοχή τους είχε μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει να το ξεχνούμε ότι όταν μιλούμε για ηλεκτρονικό εμπόριο είναι με μια τεχνολογία, αλλά πίσω από την τεχνολογία βρίσκονται και άνθρωποι και χρειαζόμαστε ανθρώπους και απευθείας διαπροσωπικές σχέσεις. Τρίτη οδηγία για τις, για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω τα σχέδια της Πολωνικής Προεδρίας για την σημαντική αυτή οδηγία που είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά αλλά και για τα επαγγελματικά προσόντα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες ό,τι αφορά την εφαρμογή την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και αυτό απαιτεί προσπάθειες όχι μόνο από τα κράτη-μέλη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ένα τομέα που έχουμε και κρατική εμπειρία. Ξέρω ότι για να εφαρμοστεί μια τέτοια οδηγία χρειάζεται να εμπλακεί ενεργά η διοίκηση. Και θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και κάποιες κρατικές ε, ιδιαιτερότητες ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανοίγματο αγοράς. Και μάλιστα έχουμε εδώ τον συνάδελφο που παρουσίασε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό για μας ε, αυτή η όθηση για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς για τις ε, υπηρεσίες να, είναι, να έχει δυναμικό χαρακτήρα. Θα στηριχτούμε και για το έργο αυτό, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στη μεθοδολογία που έχει δοκιμαστεί σε διάφορου τομεί, όπω είναι ο οικοδομικό, τουριστικό, οι υπηρεσίε για τι επιχειρήσει, που συμπεριλήφθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα στη διάρκεια τη ε, Ουγγρική Προεδρία. Εμεί δεν πρόκειται να αναλάβουμε νομοθετικέ δράσει ε, στον τομέα αυτό. Θα συνεχιστούν μόνο οι εργασίε ό,τι αφορά τη διαδικασία τη αμοιβαία αξιολόγηση στα πλαίσια της οδηγίας ε, για τους εσωτερικούς ε, για τις οδηγίες για τους υπηρεσίες ιστορικής αγοράς. Ήθελα επίσης ε, να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για την έκθεση της κυρίας Μαρκοζάτα Χάντζλικ για, τον, για το μηχανισμό αυτό αμοιβέ αξιολόγηση. Είναι ένα νεωτεριστικό εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους τομείς. Ένα τέταρτο τομέα είναι η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή δεξιοτήτων. Η Πολωνία πιστεύει μετά από ανάλυση των μέχρι τώρα προ... εμπειριών είναι ότι χρειάζεται μια τροποποίηση και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γιατί μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξεχρονισμό της οδηγίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και θα εξετάσουμε με προσοχή και την σχετική έκθεση που ετοιμάζει η κυρία Έμι Μακλάρκιν. Πέμπτο θέμα είναι η πρόταση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να καταλήξουμε σε αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των κανόνων ή των προδιαγραφών, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία σε τέτοιες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του κανονισμού παρά των οδηγιών, για να έχουμε ομοιόμορφα και νέα στάνταρ προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να έχουμε τέτοιες ομοιόμορφες προδιαγραφές, καλό θα ήταν να έχουμε κανονισμό και όχι ε, οδηγία γιατί ο κανονισμός είναι άμεση εφαρμογής, ενώ η διαδικασία για την εφαρμογή της οδηγίας είναι πιο χρονοβόρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έντβαρτ Κοζούσνικ για την έκθεσή του που προτείνει ενδιαφέρουσες συστάσεις για τη συμπλήρωση της κοινωτικής νομοθεσίας για το θέμα αυτό. Γιατί ε, η ενιαία προδιαγραφή για τους φορτωτές των κινητών είναι ίσως ε, μια συμβολική πρωτοβουλία που πραγματικά αποδεικνύει πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε μια ενιαία προδιαγραφή και πόσο θα μας διευκολύνει την καθημερινότητα αν έχουμε ένα, μια ενιαία προδιαγραφή για ενιαίο φορτωτή για τα κινητά. Επίσης, θα ήθελα να επενέσω την εισηγήτρια Λάρα Κόμη ε, που ασχολείται με την οδηγία για την εναρμόνιση των τύπων και των κανόνων. Το θέμα της ευρωπαϊκής ε, τυποποίησης είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται και φυσικά με τον τομέα των υπηρεσιών. Ένα άλλο θέμα είναι ο κανονισμός ε, για τα οχήματα με κινητήρα, τους ελκυστήρες και τα οχήματα 2, 3 ή 4 τροχών. Αυτό το θέμα για την Πολωνική Προεδρία θα είναι σημαντικό. Θα συνεχίσουμε τις προηγούμενες εργασίες ε, της Βελγικής και Ουγγρικής Προεδρίας σε στενή φυσικά συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέποντας ε, σε υιοθέτηση μιας πρότασης ε, κανονισμού για τα οχήματα αυτά. Και φυσικά και εδώ προσβλέπουμε σε στενή και επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή σας, τον κύριο Βιμ Βαντενκάμπ και τον κύριο Πιεραντώνιο Έβδομη προτεραιότητα είναι τα νομοθετικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την εισαγωγή προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσαρμογή 10 οδηγιών. Πρόκειται για τεχνική μεν, πολύ σημαντική δε ε, νομοθεσία. Γιατί θα προσαρμόσουμε 10 οδηγίες στα νέα νομοθετικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την εισαγωγή προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά αυτό το θέμα για μας είναι προτεραιότητα. Ένα άλλο θέμα αφορά την αλλαγή του κανονισμού, την τροποποίηση του κανονισμού για την περιαγωγή. Και αυτή είναι πολύ σημαντική απόφαση για τους καταναλωτές και πολύ σημαντική απόφαση για τους Ευρωπαίους για να μην έχουμε στον τομέα αυτό τόσο σημαντικούς οικονομικούς φραγμούς όπως σήμερα. Η άρση αυτών των φραγμών θα βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τέτοιος κανονισμός λοιπόν θα πρέπει να άρει τους μονοπωλιακούς τεχνικούς φραγμούς. Χρειάζεται ένας τέτοιος κανονισμός και το ξέρουν αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες, γι' αυτό τον απαιτούν. Ένατη πρωτοβουλία αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία για τις δημόσιες προμήθειες και τις συμβάσεις παραχώρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και η Πολωνική Προεδρία θα εξετάσει το σχέδιο οδηγίας που τροποποιεί την προηγούμενη οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες και μάλιστα το, την πρόταση της, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περιμένουμε τον, το νωρίτερο στα μέσα Ιουλίου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι ήδη από τον Αύγουστο γιατί σας διαβεβαιώνω ότι φέτος η Πολωνία δεν θα έχει καθόλου διακοπές, γιατί προετοιμάζουμε και τις βουλευτικές εκλογές, οπότε θα είμαστε συνεχώς σε γρήγορση, δεν πρόκειται να κάνουμε καθόλου διακοπές φέτος. Πολύ σημαντική θα είναι και η έκθεση της κυρίας Χάιντε Ρούλε, με θέμα τον εξυγχρονισμό των διατάξεων για τις δημόσιες προμήθειες. Διαβάσαμε τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής, που αφορούν κυρίως την πρόθεση της καινοτομίας και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Από αυτή την άποψη, οι δημόσιοι πόροι και οι δημόσιοι φορεί θα πρέπει να προωθούν τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Δέκατο σημείο είναι ο κανονισμό για την εκτέλεση από τι τελωνιακέ αρχέ των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα νέο κανονισμό σε ό,τι αφορά την εκτέλεση τέτοιων δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία από τι τελωνιακέ αρχέ. Αυτό εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εντάσσονται και στην ε, στρατηγική της ενιαίας αγοράς. Χαίρομαι γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο εισηγητής ε, Γιούργεν Κρόιτσμαντ ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα έχουμε στενή συνεργασία και μαζί του. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και ιδιαίτερα την, ε, την εισηγήτρια Ρούζι Τούν και τον Ανδρέα Σβάμπ καθώς και τον ε, κύριο Λούι Γκρέχ για την ε, ανάληψη της πρωτοβουλίας άνευ προηγουμένου που είναι αυτό το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς για την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς, την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών. Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα στην Κρακοβία 2 με 4 Οκτωβρίου του 2011. Η Πολωνική Προεδρία φυσικά είναι ανοιχτή και πρόθυμη για συνεργασία μαζί σας και θα είναι βέβαια οι τελευταίες μέρες της Πολωνικής Προεδρίας στις 9 Οκτωβρίου θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές, οπότε θα είναι πανηγυρικός τρόπος για την ολοκλήρωση το, της κοινοβουλευτικής μας θητείας στην Εθνική Βουλή και ελπίζω να συμβάλλουμε με το φόρουμ αυτό ε, στην προώθηση της κοινή ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ. that was quite extensive, if there will be questions. very βεβαίως και θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος, αλλά ίσως πρέπει να ακούσουμε ε, την επόμενη εισήγηση από την κυρία Κρασνοντεπεσκή, ε, που είναι αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού. Ίσως μπορείτε εσείς ε, να μας μιλήσετε λιγάκι για τα θέματα του τομέα σας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα κατά την έναρξη της Πολωνικής Προεδρίας να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για την προστασία του καταναλωτή στην ενιαία αγορά και να σας παρουσιάσω και τις ιδέες που ενέπνευσαν τις προτεραιότητες. Η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική γιατί γνωρίζω ότι για να υλοποιήσουμε μια επιτυχή προεδρία θα πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα αυτό έδειξε η εμπειρία των προηγούμενων προεδριών ότι η επιτυχής προεδρία κρίνεται από την εντατική και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γιατί το Κοινοβούλιο πραγματικά εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό συμφέρον, τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις, γι' αυτό και χρειάζεται ε, εμβάθυνση της συνεργασίας, καλύτερη συνεργασία προκειμένου να έχουμε αποτελεσματικότητα μεταξύ του κοινοτικού, του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά θα πρέπει να φανεί και ενωμένη. Μεταξύ των φραγμών που εντοπίσαμε στα, στην προστασία του καταναλωτή. Διαπιστώσαμε την έλλειψη της εμπιστοσύνη ε, στο διασυνοριακό εμπόριο, κάποια διοικητικά γραφειοκρατικά εμπόρια, νομικά, νομικά εμπόδια, το θέμα της ε, αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών και το θέμα της έρευνας των ε, αξιώσεων. Βέβαια, η υπέρβαση όλων αυτών των εμπορίων είναι σημαντικές προτεραιότητες για να ευαθύνουμε την ενιαία εσωτερική αγορά, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Παύλακ. Μόνο έτσι θα επαναφέρουμε την Ευρώπη στο δρόμο της αηφόρου ανάπτυξης. Και μάλιστα αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν θα γιορτάσουμε την 20η επέτειο των εγγενείων της εσωτερικής αγοράς. Σε ό,τι αφορά τις ε, πολωνικές προτεραιότητες θα ήθελα να επικεντρωθώ σε πέντε τομείς. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών στα έτη 2014-2020. Από αυτή την άποψη μεγάλη σημασία θα έχει η έναρξη της ε, των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπόνηση νέας στρατηγικής πολιτικής καταναλωτή για την περίοδο 2014-2020. Θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια και αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία των ασθενέστερων πλευρών της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία και από την άποψη αυτή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή σα. Ελπίζω ότι νέα αυτή η στρατηγική θα υθετήσει καινοτόμα προσέγγιση και εγκάρσια η οριζόντια προσέγγιση, ώστε να λάβει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Εύα Μπριτσπέσο που είναι συγκέντρια για το θέμα αυτό. Άλλος τομέας είναι η, η οριζόντια οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ε, βέβαια η επίσημη έγκριση τη οδηγία αυτή, ε, ελπίζω να γίνει στη διάρκεια τη Πολωνική Προεδρία μετά την διόρθωση από νομική και γλωσσική άποψη του κειμένου. Ελπίζουμε ότι τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχέ Οκτωβρίου θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτό αυτή την οδηγία και θα ήθελα να επενέσω εδώ το έργο τη Επιτροπή και τη συμβολή του Προέδρου του κ. Χάρμπορ για την προώθηση αυτών των εργασιών καθώ ε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ανδρέα Σβάμπ, τον εισηγητή που προσπάθησε τα μάλα σε αυτό το πολύχρονο και δύσκολο σχέδιο. Επόμενη προτεραιότητα αφορά τον εναλλακτικό τρόπο διακανονισμού των διαφορών. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες και στον τομέα αυτό με την πρωτοβουλία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποβληθούν κάποια σχέδια σε ό,τι αφορά τον εναλλακτικό μηχανισμό διακανονισμού των διαφορών, ADR, και ταυτόχρονα ε, online επίλυσης διαφορών, ODER, επιγραμμικής επίλυσης διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει, θέλει να καταστήσει πιο αποτελεσματικά τα διάφορα όργανα ε, διακανονισμού των διαφόρων με βάση το, την ανακοίνωση για το Single Market Act και μάλιστα το ADR, αυτή η εναλλακτική επίλυση των διαφορών, είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί συμφωνούμε με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι μηχανισμοί διακανονισμοί των διαφορών θα πρέπει να είναι εύκολοι, φτηνοί, απλοί και εύκολη πρόσβαση για τους καταναλωτές και μεγάλο πλεονέκτημα του ADR είναι η ελαστικότητά του. Ε, μπορεί να γίνεται ελαστική επιλογή ανάλογα με το είδος της διαφοράς. Έτσι θα μειωθούν και οι επιβαρύσεις στο δικαστικό σύστημα. Και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία για τον ελεκτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών συνοδεύεται από την online επίλυση των διαφορών, το OIDR, και εδώ μπορούν να διαλευκανθούν κάποιες διαφιλονικίες ό,τι αφορά διασυνοριακές συναλλαγές. Και μάλιστα η πρόθεση αυτών των δύο πρωτοβουλειών είναι σημαντική για την πολιτική προστασία του καταναλωτή. Α μην ξεχνούμε και την ανάγκη διαπαιδαγώγηση και ενημερωτική εκστρατεία που θα πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό, για να είναι αποτελεσματικοί οι δύο μηχανισμοί επίλυση των διαφορών. Επίση, θα πρέπει να προβλέψουμε και κάποιε νομικέ διατάξει για να εξασφαλίσουμε και την πρόθεση τη διαιτητική ε, επίλυση των διαφορών. Νομίζω ότι ε, πολλές φορές η χαμηλή πρόσβαση στην διαιτησία οφείλεται στην άγνοια των φορέων της αγοράς. Αυτό έδειξαν και οι πρόσφατες διαβουλεύσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πολωνική Προεδρία θα υποστηρίξει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να θεσπιστεί ένας κοινοτικό μηχανισμός εναλλακτικού διακανονισμού των διαφορών και προσβλέπουμε και εδώ σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και με τον αρμόδιο συγκητή, τον κύριο Ρομπέρ Ροσφόρ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μετά την υποβολή της επίσημης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενος τομέας είναι η αναμενόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την οργάνωση ε, διακοπών, εκδρομών και ταξιδιών. Αυτό το package travel είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της αγοράς και ο τουρισμός αυτή τη στιγμή πλήττεται γιατί υπάρχουν κάποια νομοθετικά κενά και δεν έχουμε αρκετές σύγχρονες διατάξεις που να επιτρέπουν τους φορείς να λειτουργούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό μεταξύ των σημαντικών ε, αιτίων της αναθεώρησης της οδηγίας που αναμένουμε είναι ο αναγκαίος εξυγχρονισμός των σχετικών διατάξεων προκειμένου να καλυφθούν τα νομικά κενά, να γίνουν κάποιες απλουστεύσεις της διαδικασίας και να αρθούν οι υπάρχοντες φραγμοί στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να έχουμε μια πιο ομοιόμορφη διαδικασία στα κράτη-μέλη. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταφέρει να υποβάλει αυτή την πρόταση στη διάρκεια της Πολωνική Προεδρίας, εκφράζουμε την ελπίδα ότι η έναρξη των εργασιών θα αποτελέσει προτεραιότητα το, του τρίου των Προεδριών με συμμετοχή της Δανίας και της Κύπρου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αναθεώρηση οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Όπω μα είπε και ο το θέμα τη εποπτεία αγορά είναι πολύ προσφυλέ για μας και μάλιστα με την ενίσχυση της ασφάλειας και της εποπτείας της αγοράς για ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουμε μια πιο ισχυρή εσωτερική αγορά. Θέλουμε να γίνει μια εξορρόπηση μεταξύ των εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ε, στοιχείων, έχοντα υπόψη τη διαφάνεια αλλά και την ανάγκη προστασία του καταναλωτή. Γι' αυτό και η Πολωνική Προεδρία θα, ξεκινήσει εργασίε με βάση το, την πρόταση αναθεώρηση οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Περιμένουμε φυσικά το σχέδιο αναθεώρησης ε, αυτής της οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως φάνηκε και από το ψήφισμα της 8ης Μαρτίου για την οδηγία της γενικής ασφάλειας των προϊόντων. Η Πολωνική Προεδρία συμφωνεί με την ανάγκη αναθεώρηση της οδηγίας για την γενική ασφάλεια των προϊόντων και περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξεκινήσουμε και εμείς τις εργασίες μας. Επαναλαμβάνω, αν η πρόταση της Επιτροπής δεν υποβληθεί στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, ελπίζω τουλάχιστον οι επόμενες Προεδρίες να θεωρήσουν αυτό το σημείο ως προτεραιότητα. Το τρίο των Προεδριών να συνεχίσει αυτό το θέμα. Θα ήθελα τέλος να υπογραμμίσω ότι μια αποτελεσματική πολιτική προστασία του καταναλωτή βελτιώνει την καθημερινότητα και τη ζωή του πολίτη καλά ενημερωμένο ε, καταναλωτή ε, που έχει συνείδηση των δικαιωμάτων του είναι κινητήριο δύναμη τη αγορά και μέχρι στιγμή αυτό το δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρω. Εμεί ε, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα του καταναλωτή και μάλιστα σε όσο δυνατό πιο πρόωρη φάση και σε αυτό προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΙΜΚΟ αλλά φυσικά ζητούμε την στήριξη και των άλλων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών και η επιτυχία τη Πολωνική προεδρία είναι επιτυχία για όλου. Θα ήθελα επίση να ευχαριστώ το προηγούμενο τρίο των Προεδριών για τι προσπάθειε του και για τι προκλήσει, τι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν στη δύσκολη αυτή περίοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και ιδιαίτερα να επενέσω την προκάτοχο Ουγγρική Προεδρία που κυρίω έφτασε σε αίσιο πέρα στην οδηγία για την προστασία του καταναλωτή θα ήθελα να σας προκαλέσω στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής ημέρας ανταγωνιστικότητας και καταναλωτή που θα γίνει στις 24 και 25 Νοεμβρίου στο Πόσμα. Αυτή η διεθνής διάσκεψη θα γίνει σε συνεργασία με τα αντιμονοπολιακά γραφεία και γραφεία προστασίας του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναλύσουμε διάφορες διατάξεις αντιμονοπολιακής νομοθεσίας και, και νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή. Είναι σημαντική η σχέση ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή και κέρια για την εσωτερική αγορά. Επαναλαμβάνω, ελπίζω να είναι ε, σημαντική και η διεθνή συνεργασία. Γι' αυτό και θα προσκαλέσουμε στη διάσκεψη αυτή τη διεθνή, αυτή τη διάσκεψη στο Πόζναν και του εταίρου μα από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε απορία σα. Well, I want to thank... Um, ευχαριστώ και τον κύριο Παύλακ και την κυρία Κρασνοντέμψκα. Βλέπετε πόση δουλειά έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ επίσης γιατί εκφράσατε την ευγνωμοσύνη σας προς όλους τους εισηγητές που εργάστηκαν τόσο σκληρά. Αναφέρατε και την Ουγγρική Προεδρία. Θέλω και εγώ να αναγνωρίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία αντιπροσωπεύεται εδώ επίσης η κυρία Γκέτεσου. που ασχολήθηκε με την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε μισή ώρα για ερωταπαντήσεις. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους εισηγητάς. Πώς θέλετε, τρεις-τρεις τις ερωτήσεις. Τρεις-τρεις. Αλλά παρακαλώ να είναι περιεκτικές και συνοπτικές οι ερωτήσεις. Ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Παύλα, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, εισήγησή σας και δείξατε ότι έχετε προετοιμαστεί θαυμάσια και για την ε, πολιτική Προεδρία και για τις εργασίες Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κ. Στούσκα, ο πρωθυπουργό σα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο έκανε μια εντυπωσιακή ομιλία για την Ευρώπη και για τι ευκαιρίε που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για μια Ευρώπη που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δυσκολίε. Ελπίζω λοιπόν κατά τους επόμενους ε, μήνες ε, να ε, συνεχιστεί αυτή η πολιτική με μεγάλη επιτυχία. Ε, θέλουμε όλοι να εφαρμόσουμε την κοινή αγορά και η Πολωνία και εσείς αναφέρετε μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην Επιτροπή μας και τα παρακολουθείτε. Και ρωτώ, Υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέμα που σας ε, απασχολεί. Εμένα που με ενδιαφέρουν οι συμβάσει παραχώρησης. Γιατί από ό,τι γνωρίζω στην Πολωνία δεν είναι ιδιαίτερα διαδομένες οι συμβάσει παραχώρησης σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχει κάποια ειδική δυσκολία για την ε, Πολωνία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας. Μετά, ψηφιακή εσωτερική αγορά. Θέλετε να την επεκτείνετε. Και εδώ ρωτώ, πώς προτίθεστε να πιέσετε την Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις. Τρίτη μου ερώτηση αφορά την κυρία Τόμπιλ από το Γραφείο για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Ανταγωνισμό και σας ερωτώ συγκεκριμένα το εξής. Υπάρχει μία πρόταση για εναλλακτική διευθέτηση διαφορών, ε, μία πρόταση κομισιών που θα κατατεθεί ε, το Σεπτέμβρη και αυτή μπορεί να ε, επικαλυφθεί εν μέρη και με την οδηγία ή την πρόταση για συλλογικές προσφυγές εσείς ε, όσον αφορά τις ε, συλλογικές ε, προσφυγές. Τι πιστεύετε. Σήμερα στην Επιτροπή μας καταλήξαμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μόνο αν αυτή η διαδικασία στηριχθεί από τα κράτη-μέλη και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μην επικρατήσουν στην Ευρώπη αμερικανικές συνθήκες. Uh, thank you, Κύριε κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία, να ευχαριστήσω εσάς ε, κύριε Παύλακ ε, για την ε, πραγματικά ευρωπαϊκή σκέψη που παρουσιάσατε. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα η πρώτη σας ε, πρόταση όπου είπατε ότι στην Ευρώπη ο σημαντικότερος στόχος είναι η ολοκλήρωση. Ε, και αυτός είναι και ο σημαντικότερος στόχος της δικής σας της πολιτικής. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα θετικό θέμα που πολλές άλλες προεδρίες δεν το ανέφεραν, το παρέλειψαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά γι' αυτό και θέλω να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, οδηγία παροχής ε, υπηρεσιών και επαγγελματικά προσόντα. Τα αναφέρατε όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικά. Όμως, ερωτώ γιατί δεν το είπατε. Αυτή η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας. Τι πιστεύετε για αυτήν έτσι ώστε οι πτυχιούχοι ε, με μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο θέμα, θίξατε το θέμα της περιαγωγής. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και επιθυμώ ε, να πω το εξής. Μήπως ε, θα έπρεπε να προχωρήσουμε περισσότερο στη συζήτηση εκεί όπου γίνεται λόγος ε, για την ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την κατάτμιση της αγοράς για να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τους πολίτες. Έχω κατά νου, ε, πολυεθνικές εταιρείες ε, οι οποίες όμως εκμεταλλεύονται αυτή την κατάτμιση της ευρωπαϊκής αγοράς και διερωτάται κανείς ε, γιατί να χρειαζόμαστε τέλη περιαγωγής τη στιγμή που πρόκειται για δύο θηγατρικές επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου η τρίτη ερώτηση προς ε, την πρόεδρο του Γραφείου Ανταγωνισμού, συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά το όνομά σας, είπατε ότι η παρακολούθηση της αγοράς είναι πολύ σημαντική και έχετε δίκιο στον τομέα της επιτήρησης ή παρακολούθησης της αγοράς υπάρχει μήπως ένας τομέας ε, που ε, να σας ε, απασχολεί ιδιαίτερα ίσως οι, οργανω... η καταναλωτών που δεν τις αναφέρετε όμως. Στην Πολωνία υπάρχουν αυτές οι ενώσεις καταναλωτών και εσείς η κυβέρνηση στηρίζετε τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτή για να μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκπληρώνουν καλύτερα τα καθήκοντά συμφέροντά τους. Then, uh, Mr. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εσάς ε, κύριε Παύλακ ε, για τα ευεργετικά σας λόγια. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω συναδέλφους ε, στη Βαρσοβία και στην Κρακοβία και μου άρεσε πάρα πολύ εμένα που είμαι Γερμανός το πώς εσείς προάγετε την κοινή αγορά. Όχι μόνο τη στηρίζετε αλλά είστε και κινητήρια δύναμη για την Ευρώπη. Το είπε και η κυρία Κέπχαρτ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και επιφυλάξει απέναντι στην Ευρώπη. Άκουσα ότι όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς είσαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Θεσμοί όπως είναι η Solvit και πολλοί άλλοι ε, στηρίζονται από εσάς και όχι μόνο αυτό αλλά έχουν και συγκεκριμένα καθήκοντα, χρησιμοποιούνται. Και εγώ έχω ερώτηση γιατί και άλλοι είχαν ερωτήσεις. Έμαθα ε, στο διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τη Γερουσία ότι εσείς ως κυβέρνηση ενδιαφέρεστε να υπάρχει ε, μια κοινή αγορά για πίστη, για δάνεια. Ε, γιατί πολλές φορές οι Πολωνοί που χρειάζονται ε, στεγαστική πίστη καταφεύγουν στο εξωτερικό, στην Ελβετία και αυτό κρίνεται ως παρεμπόδιση της κοινή αγοράς. Θυμάμαι που είπατε ότι αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τους Πολωνούς γερουσιαστές. Δεν τους αρέσει και το κατανοώ ότι για σας θα ήταν πρόοδος για αυτό το θέμα να αλλάξει η κοινή αγορά. Κατά τα άλλα σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε η κινητήρια δύναμη για την ε, κοινή αγορά και όχι μόνο για την ολοκλήρωση της κοινή αγοράς αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης. Επιθυμείτε παρακαλώ να απαντήσετε σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Απευθύνομαι και στους ε, δύο μιλητές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, για τους μηχανισμούς που θα στηρίξουν την εσωτερική αγορά, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη σωστής στάθμισης ε, της νομοθεσίας. Αυτό που απαιτεί η νομοθεσία θα πρέπει να είναι σωστό. Δεν θέλουμε μόνο ευνομοθετήν, αλλά και έξυπνο νομοθετή. Θέλουμε έξυπνη, εύστροφη νομοθετική διάταξη. Και επίσης θέλουμε να περιορίσουμε το διοικητικό φόρτο, το γραφειοκρατικό άχθος και τις ε, πληροφορίες, τις υποχρεώσεις ε, πληροφόρησης. και διαπίστωσα ότι πολύ συχνά η διοίκηση έχει μία τάση να οχυρώνεται πίσω από τις θέσεις της. Τώρα προσπαθούμε να περιορίσουμε τις απαιτήσει για, ε, για την ενημέρωση και να ε, γενικεύσουμε τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων που αντικαθιστούν τα γραπτά. Αλλά αυτό δεν γίνεται τελικά, είναι ανέφικτο. Δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα που δεν μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την πρόταση. Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή αγορά και ποιες είναι οι προσδοκίες για την ψηφιακή αγορά, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στα ζητήματα τα σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή. Θα πρέπει και εδώ να έχουμε διαφανείς προδιαγραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι σήμερα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι χρήσιμη μια τέτοια συζήτηση. Και εδώ έρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Γκέπχαρτ για την περιαγωγή. Χρειάζεται μία συζήτηση για την κατάσταση αυτή και για την ενημέρωση. Έχουμε πολύ σημαντικό βιβλίο, το The Master Switch. Και μάλιστα το βιβλίο αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η, και πόσο αναγκαία είναι η εφαρμογή παρόμοιων κανόνων σε όλη την ε, ε, ενεργειακή αγορά, ώστε όποιος παράγει την πληροφορία να μην έχει το ε, μονοπόλιο ούτε στην, με, ούτε στην μεταποίηση της πληροφορίες είτε στην απόσυρση της πληροφορία. για να μην ε, ε, δημιουργείται ε, κυρίαρχη θέση αυτού που παράγει την πληροφορία. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίσουμε, να εκπονήσουμε κάποιους μηχανισμούς ώστε να υπάρχει μια, ένα σωστός διαχωρισμός για να αποφευθούν τα μονοπόλια. Οπότε σημαντική είναι η συζήτηση για το πώς λειτουργεί η σύγχρονη κοινωνία, ε, μια κοινωνία στην οποία η πληροφορία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να μην γίνουμε όμοιροι ή εχμάλωτοι κάποιων τεχνολογιών και κάποιων ε, μηχανισμών. Να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα ε, πρόσβασης και νέων επιχειρήσεων στην αγορά, υποβολής και νέων ιδεών στην αγορά, να μην υπάρχει ένα περιορισμένος χώρος. Και το θέμα της περιαγωγής είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να είμαστε και πιο φιλόδοξοι, να έχουμε περισσότερη πρόοδο. Φυσικά, φυσικά, μπορούμε. Στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει roaming, δεν υπάρχει περιαγωγή, οπότε είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σταδιακή προσέγγιση. Να μην βιαστούμε, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε προβλήματα και στις επιχειρήσεις. Γιατί αν έκαναν τις επενδύσεις τους με διαφορετικό μοντέλο, αν υιοθέτησε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο με συγκεκριμένες διατάξεις, δεν μπορούμε ξαφνικά να αλλάζουμε το τοπίο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις α, ε, ρυθμίσεις, τις διατάξεις που ανέφερε ο κ. Κρόισμαν, το μηχανισμό Solvit είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός στήριξης των επιχειρήσεων και αυτό που είναι σημαντικό στις α, ε, υπηρεσίες πληροφορίας είναι να προωθήσουμε ταυτόχρονα την πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ε, όταν προσθέσουμε τα κινέζικα ή τα ιαπωνικά έχουμε μόνο μία στήλη στην βάση δεδομένων, οπότε αυτή την άποψη ε, θα έχουμε ήδη παγκόσμιες υπηρεσίες. Ε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην πολυγλωσία και φυσικά στην προεργασία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις, τα δάνεια που συνάπτονται με ρήτρα συναλλάγματο, αυτό είναι μάλλον εσωτερικό πρόβλημα τη Πολωνία. Μερικές χώρες έχουν πληγεί γιατί με την αλλαγή της ισοτιμίας βρέθηκαν σε πολύ δυσμενή θέση όσοι έχουν τέτοια δάνεια με ρήτρα συναλλάγματος. Εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει σε τέτοιο είδους δάνειο κίνδυνος της αλλαγής εναλλαγματικής οτιμίας και στην Πολωνία οι τράπεζες ε, είχαν μεγάλο spread, υιοθέτησαν μεγάλο spread μεταξύ αγοράς και πώληση και στα ενυπόθηκα δάνεια έχουν, υιοθετούν spread πάνω από 20%. Ε, συγγνώμη, 12%. Ε, είναι σημαντικό αυτό, ε, αλλά γίνεται η αναγραφή άμεσα σε συνάλλαγμα. Και νομίζω ότι αυτός ο μηχανισμός είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός ανταγωνισμού. Αν οι τράπεζες δεν, δεν θέλουν να πωλήσουν συνάλλαγμα με λογική τιμή, ο πελάτης μπορεί να διαλέξει να αγοράσει συνάλλαγμα σε άλλη τράπεζα ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα να αποτανθεί διαφορετικά για να αναγκάσει τις τράπεζες να μειώσουν αυτό το spread συναλλάγματος. Η μείωση αυτού του spread θα είναι επωφελής και για τους πελάτες. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σήμερα ότι σήμερα οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ε, επηρεάζουν πολλές φορές την ανταγωνιστικότητα. Και βλέπετε τη σχέση συναλλαγματικής ισοτιμίας και ανεργίας. Στις αρχές της δεκαετίας, όταν για ένα ευρώ μπορούσαμε να πληρώσουμε 90 ε, cent αμερικανικά, η ανεργία τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, χαμηλότερη από τη σήμερα. Όταν ενισχύθηκε το ευρώ, όταν ε, άλλαξε η συναλλαγματική ισοτιμία και όταν ένα ευρώ ήταν 1,60 δολάρια, τότε αυξήθηκε και η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι είναι ελληνέντατα τα θέματα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή της συναλλαγματικής πολιτικής και της απασχόλησης, γιατί η συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και άρα τη δημιουργία ή την απώλεια θέσεων απασχόληση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, νομίζω ότι είχατε και εσείς μερικά θέματα. Ευχαριστώ. Όντως έγιναν ερωτήσεις και για θέματα πολιτικής καταναλωτών. Ε, η πολιτική καταναλωτών είναι πολύ σημαντική για μας ε, στην Πολωνική Προεδρία. Ο κύριο Φαβ ε, μίλησε για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και τις συλλογικέ προσφυγές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί αφορά την ενίσχυση της εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην αγορά. Επίσης και αυτό το θέμα ενδιαφέρει την Επιτροπή ΙΜΚΟ και εξετάσουμε τις λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, μεταξύ των δύο συστημάτων. Το ADR, αναλλακτικός μηχανισμός, ε, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βρίσκεται ε, στο, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων ήδη στη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας και μάλιστα υπάρχει ένα έγγραφο που μιλά για τους σημαντικούς μοχλούς που είναι οι μηχανισμοί αυτοί στην ενιαία αγορά και γι' αυτό υπάρχει δέσμευση και η ετοιμότητα της Πολωνικής Προεδρίας να προωθήσει το έγγραφο αυτό για τον εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Βέβαια για να γίνει δυνατή η έναρξη των εργασιών είναι η υποβολή του, της νομοθετικής πρότασης. Τώρα σε ό,τι αφορά το σχέδιο για τις συλλογικές προσφυγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη εργασίες, ούτε έχει διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο για τις συλλογικέ πρόσφυγες. Η Πολωνική ε, Προεδρία είναι υπέρ της διευκόλυνσης των καταναλωτών και της διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να εξυπηρετούν τις ε, απαιτήσει, τους αξιώσεις τους ε, με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και κατά του αθέμητου ανταγωνισμού. Εμείς είμαστε υπέρ τέτοιων μηχανισμών που φυσικά δεν ε, θα διευρύνει απλώς το αμερικανικό μοντέλο, αλλά θα προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες, θα είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο και θα λαμβάνει υπόψη τις δικές μας ιδιαιτερότητες, τις δικές μας νομικές παραδόσεις, αλλά και τη, την ε, ισχυρή νομική και διοικητική ε, ρύθμιση που ισχύει σε διάφορες χώρες, ειδικά και στην Πολωνία. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει τη κυρία Γκέπχαρτ για την εποπτεία τη αγορά και την, το ρόλο των οργανώσεων καταναλωτή, το θέμα αυτό μα είναι ιδιαίτερα προσφυλέ. Και φυσικά εγώ είμαι πρόεδρος ε, του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή. Το πολωνικό σύστημα περιλαμβάνει πολλά θεσμικά όργανα ε, και η κρατική πολιτική για την προστασία του καταναλωτή προβλέπει υποστήριξη τέτοιων οργανώσεων και μάλιστα έχουμε ήδη μια στρατηγική μέχρι τα τέλη του 2013 μα το έγγραφο που δώσαμε έτυχε της υποστήριξης της πολωνικής κυβέρνησης και μπορώ να σας δώσω αυτό το έγγραφο και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό που προβλέπει στήριξη του ανταγωνισμού, του ανοιχτού ανταγωνισμού και της ενίσχυσης της οργάνωσης ε, προστασίας του, των οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή, γιατί το γραφείο μας έχει δύο αρμοδιότητες, και τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή. Θέλουμε λοιπόν και ισχυρές οργανώσεις καταναλωτή, αλλά και ισχυρό ανταγωνισμό. Θέλουμε καλή θέση για τις οργανώσεις του καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των κρατικών κονδύλιων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω 12 εγγεγραμμένους και μόνο 20 λεπτά. Ίσως να παίρνουμε τις ερωτήσεις 4-4. Ο κύριος Μπίλαν ήταν στην προηγούμενη φορά ο τελευταίος συντονιστής που μίλησε. Ο κύριος Μπιέλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Γενική Διευθύντρια. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Βέβαια με τον ε, Προεδρεύοντα είναι η δεύτερη συνάντηση. Συναντηθήκαμε στην ομάδα των συντονιστών την πρώτη φορά και εκεί αναλύσαμε και πάλι το πρόγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας. Ε, χαίρομαι για το ότι λάβατε υπόψη και κάποιες παρατηρήσεις που κάναμε τότε συνεδρίαση με τους συντονιστές. Είπατε ότι η Πολωνία είναι θερμός υποστηρικτής της εσωτερικής αγοράς και θέλει να γίνει ο πρέσβης της εσωτερικής αγοράς στο επόμενο εξάμεινο και αυτό φαίνεται με την ανάλυση των προτεραιοτήτων της Πολωνικής Προεδρίας και την ανάλυση των του προγράμματος των διαφόρων εκδηλώσεων. Θα είναι οργανώτρια της Ευρωπαϊκής ημέρας ε, ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή, θα οργανώσει το πρώτο φόρουμ εσωτερικής αγοράς. Έχω μόνο δύο παρατηρήσεις, δεν θα ήθελα να γίνει πολλών πολωνική συζήτηση. Έχω δύο παρατηρήσεις και μία ερώτηση. Το πρόγραμμα της πολωνικής προεδρίας είναι υπερβολικά φιλόδοξο, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι και εφικτό και θα προλάβετε να, θα προλάβετε να το εφαρμόσετε. Ειδικά για την οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, οι Πολωνοί οι ευρωβουλευτές έδωσαν μάχη πραγματικά ε, και έκαναν μεγάλες προσπάθειες. Τελικά δεν μείναμε ικανοποιημένοι από, δεν μείναμε ικανοποιημένοι το Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ε, το χρονοδιάγραμμα της Πολωνικής Προεδρίας θα συμπέσει με την προεκλογική σας εκστρατεία και ο Πρωθυπουργός είναι και αρχικός του κόμματός σας. Οπότε θα απασχοληθεί και με τα προεκλογικά ζητήματα. Ελπίζω σε μισό χρόνο, σε ένα εξάμεινο που θα ξανασυναντηθούμε, να κάνουμε ένα θετικό απολογισμό της Πολωνικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που επισήμανε η κυρία Γκέπχαρτ, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην περιαγωγή. Γιατί ε, πραγματικά είναι ένα χαράτσι ε, αυτό που επιβάλλεται στα τέλη της περιαγωγής. Έχουμε ε, στην Πολωνία γαλλικές ε, εταιρείες, στην Orange ή τη γερμανική στην T-Mobile που αγοράζουν τοπικούς ε, παρόχους υπηρεσιών και επιβάλλουν τα τέλη που θέλουν. Είναι πραγματικά ένα χαράτσι αυτό που πληρώνουν οι χρήστες εξαιτία της περιαγωγής. Είπατε ότι θέλετε σταδιακή προσέγγιση. Το ίδιο κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο προηγούμενος κανονισμός ήταν από το 2007 Ήδη έχει περάσει πολλής χρόνος και πολύ αργά είναι τα βήματά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει η πολωνική κυβέρνηση με πιο επιθετικό τρόπο να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλει προτάσεις. Ο κύριος Ξίστοφ Καβιατχόσκη, ο Πολωνός υπουργό Δικαιοσύνης, στα πλαίσια των εγγενείων της Πολωνικής Προεδρίας, είπε ότι θα προσπαθήσει να επιφέρει την, το, το γαλάζιο αυτό αποτύπωμα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ελπίζω να υπάρχει συντονισμός και με σας ε, κύριε Παύλα και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όντως υπάρχει ε, συντονισμός και συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν ε, και άλλους, αλλά αν έχετε καλοσύνη από μία ερώτηση ο καθένας, γιατί τελείως δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Θα μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουν όλοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις που επιθυμούν. Η κυρία Τόμκελ είπε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είναι πλήρως κατατοπισμένοι ή αγνοούν τα δικαιώματά τους και έτσι δεν μπορούν πλήρως να ασκήσουν τα δικαιώματα συμμετοχής στην εσωτερική αγορά. Η πολωνική, αγορά, η πολωνική συγγνώμη, προεδρία επικεντρώνεται στην εσωτερική αγορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και Ελπίζω να συμβάλλει η Πολωνική Προεδρία στην ενημέρωση των καταναλωτών, στην συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων τους για να μπορούν να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους και να απολαύσουν πραγματικά την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό οργανώνουμε άλλωστε και το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την ε, αφύπνιση κατά κάποιο τρόπο των Ευρωπαίων πολιτών. Και έχω και μία ε, ερώτηση. Θέλουμε περισσότερη δέσμευση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο Πρωθυπουργό Τούσκ μίλησε για περισσότερη Ευρώπη. Πώς θα το κάνουμε όμως, η εσωτερική αγορά είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, θέλουμε συγκεκριμένες λύσεις για συγκεκριμέ... που να δίνουν στους καταναλωτές την αίσθηση ότι πραγματικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Έχουμε μία σαφή, ορατή, απτή προτεραιότητα σε αυτή να επικεντρωθούμε ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ότι να, έκανε κάτι για μένα η Ένωση. Σήμερα μιλάμε για την περιαγωγή. Πραγματικά, αυτό είναι ένα θέμα που βασανίζει τους πολίτες, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, η Ευρώπη χωρίς σύνορα, η Ένωση χωρίς σύνορα στην Πολωνία. Και πολύ συχνά οι πολίτες λένε αυτό που με ενοχλεί, αυτό που με βασανίζει είναι το roaming στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορώ να έχω προσιτές ε, τιμές για τις ε, υπηρεσίες του Ιντερνετ θα μπορούσε η περιαγωγή να είναι ένα συγκεκριμένο αυτό σχέδιο για να καταλάβει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή για μας γιατί έκανε το α, το β για να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ κυρία Σαλντεμόζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Πολωνική Προεδρία που είναι τόσο δεσμευμένη για την προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά και ένας τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εδώ και καιρό είναι η ασφάλεια των προϊόντων και η επιτήρηση της αγοράς, η υποπτία της αγοράς. Ίσως δικαίως δεν υπάρχει μεγάλη πίστη στην εσωτερική αγορά γιατί πολλές χώρες έχουν περικόψει τους προϋπολογισμούς τους ή τα κονδύλια τους που αφιέρωναν προηγουμένως στην εποπτεία της αγοράς και στην προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να τις πείσουμε και αυτές ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τον έλεγχο της εσωτερικής αγοράς. Είναι κάτι ουσιώδες αν θέλουμε να επανέλθει η αξιοπιστία στους πολίτες προς την εσωτερική αγορά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ την Πολωνική Προεδρία πρώτον διότι ο καθένας μας έλαβε ένα γράμμα με τις τρεις κύριες προτεραιότητες την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δηλαδή με αναπτυξιακή διάσταση. Έπειτα Μα στείλατε ένα who's χους-χου με όλες τις σημαντικές προσωπικότητες των Υπουργείων που μπορούμε, με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε σε επαφή γραπτός. Αυτό είναι πρωτότυπο και ασυνήθιστο και πολύ θετικό. Τώρα, με βάση τις τρεις προτεραιότητες που αναφέρατε, θέλω να μιλήσω για τον προϋπολογισμό ως βασική πρόκληση της Προεδρίας σας γιατί μπαίνουμε τώρα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στο Συμβούλιο. Γνωρίζετε ότι το, Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό συζητάει τον προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό αυτό λέτε, τον προϋπολογισμό αυτό λέτε ότι θέλετε να τον στρέψετε προς τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει και δημόσιες αγορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε σε αυτές τις δημόσιες αγορές, την προστασία της καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσες είναι σε θέση να το κάνουν, αλλά που αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται έπειτα. Ως τρίτη προτεραιότητα μιλήσατε για εταιρική σχέση προς την Ανατολή και προς τον Νότο για περισσότερο εκδημοκρατισμό, για νέες αγορές με τους εταίρους αυτούς. Και υπάρχει το θέμα της αμοιβαιότητας που τίθεται. Ξέρω ότι έχετε και εσείς προβλήματα με ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα με την Κίνα. Και αυτό συζητιέται πολύ από την, στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Πώς σκοπεύετε να το θίξετε στο Συμβούλιο ώστε να πετύχουμε νέες αγορές και προς την Ανατολή. Για την επαγγελματική κάρτα μίλησε η Ευελίνα, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα ενδυναμώνατε το σύστημα IMI ώστε να επανέλθει η αξιοπιστία στους καταναλωτές και καταναλώτριες ιδιαίτερα επειδή εσείς κυρία μου ασχολείστε με τους καταναλωτές τους πιο ευάλωτους από αυτούς, τους πιο αδύνατους πώς θα τους προστατεύσετε. Τέσσερα ερωτήματα μαζεμένα. Αλλά αφού είστε αντιπρόεδρος, για να ακούσουμε λοιπόν τις απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση, η παρατήρηση μάλλον, αναφέρθηκε στον υπερβολικά φιλόδοξο χαρακτήρα του προγράμματος ε, της Πολωνικής Προεδρίας. Θα καταφέρουμε κύριε Ευρωβουλευτά, ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συνδυασμό με την προεκλογική εκστρατεία για τι βουλευτικέ εκλογές, η Πολωνική Προεδρία είχε προγραμματιστεί πολύ νωρίτερα, στα μέσα της κοινοβουλευτικής αιτία. Και μάλιστα όταν εσείς συμμετείχατε στην ε, στο κυβερνητικό συνασπισμό χάρη σε εσά ε, περιορίστηκε, συρρυκνώθηκε η κοινοβουλευτική θητεία. Εσεί μα υποχρεώσατε να, ε, βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να, συμπίπτει η Προεδρία με τι ε, προεκλογέ. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται τα δύο θέματα, αλλά η προεκλογική εκστρατεία άλλο η Πολωνική Προεδρία. Άλλωστε η εθνική εκστρατεία, η εθνική προεκλογική εκστρατεία είναι πάντα φλέγουσα, οι συζητήσει είναι σε αυτό δεν το αποφεύγουμε. Τώρα ως προς την περιαγωγή. Συμφωνώ ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολύ περισσότερες πιέσεις για διαθέτηση και όπως είπατε και εσείς κύριε Μπιεράν, αν βρούμε λύσεις στην περιαγωγή θα έχουμε πραγματικά ένα απτό αποτέλεσμα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί, για παράδειγμα, το Σέγγεν και η ελεύθερη διακίνηση ε, έχει γίνει πια δεδομένο για τους πολίτες. Ε, δεν υπάρχουν βίζες, δεν υπάρχουν προβλήματα, έχουν ήδη συνηθίσει, αλλά μερικές φορές ε, οι λύσεις είναι πολύ πιο προοδευτικές και θέλουμε να έχουμε βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και στα πλαίσια αυτά εξετάζουμε και τις ρυθμίσεις για, το, για την περιαγωγή. Δεν είναι μόνο η περιαγωγή, έχουμε και άλλους τομείς. Πάντως προσπαθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα γενικό πλαίσιο και η Πολωνική Προεδρία αλλά και εγώ προσωπικά πιστεύουμε στην ανάγκη σωστής πρώτα διάγνωσης για το τι χρήζει κοινοτική ρύθμισης και τι, σε τι τομέα θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση. Γιατί για μερικά θέματα θέλουμε ε, γενική, κοινοτική και ομοιόμορφη ε, ρύθμιση, αλλά μερικές φορές οι επιχειρηματίες παραπονούνται γιατί η υπερβολική ρύθμιση μερικές φορές είναι περίτη και η υπερβολική ομοιοπορφοποίηση. Σε ό,τι αφορά την γαλάζια αυτή, το, τη γαλάζια σφραγίδα, το γαλάζιο αποτύπωμα που ανέφερε ο Υπουργό Δικαιοσύνη, θα δώσω το λόγο στην κυρία Τόμκιλ γι' αυτό. Ένα άλλο σημείο ε, που ανέφερε μια Ευρωβουλευτή είναι να έχουμε ε, ρυθμίσεις που είναι ορατές για τον πολίτη. Για παράδειγμα, η σχέση παραγωγών και δικτύων διανομής. Και σίγουρα καλό θα είναι σε αυτή την κοινωνικό, οικονομική συνεργασία να έχουμε σωστές ρυθμίσεις, γιατί σε εμά τα δίκτυα διανομής ε, επιβάλλουν στους προμηθευτές πολλά και διάφορα τέλη για τη διαφήμιση, για την επέτειο του σούπερ μάρκετ, για πολλές και διάφορες ε, περιστάσεις. Και αυτό κάπως ε, ε, επισκιάζει τα πράγματα και δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματική τιμή, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους και αυτό δημιουργεί κνευρισμό στους παραγωγούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ρυθμίσεις που να δημιουργούν πλαίσιο για καλή συνεργασία για να μην απογοητεύσει η εσωτερική αγορά γιατί είχαμε πριν από δύο χρόνια ξεκινήσει τον κώδικα βέλτιστων των πρακτικών. Αλλά δυστυχώς δεν απέφερε καρπούς και στην οικονομική πρακτική αλλά και στην ομολογία είδαμε ότι δημιουργήθηκαν διάφορα προηγούμενα και δεδικασμένα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των προμηθευτών και των δικτύων διανομής. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα γενικό πλαίσιο για να ρυθμίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά πολλές φορές οι φορείς της αγοράς, ε, λαμβάνοντας υπόψη το, διάφο, το διαφορετικό συσχετισμό δυνάμεων, δεν είναι πρόθυμοι για συμφωνία ε, για το πού χρειάζεται ρύθμιση και πού η ρύθμιση είναι περίτη για να εξασφαλιστούν αγαστές σχέσεις. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων... Α, συγγνώμη, ξέχασα μια άλλη ερώτηση της κυρίας Σαλντεμόζε για την ενίσχυση της εποπτείας. Είπατε ότι χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία ελέγχου και εποπτείας, αλλά μερικές φορές ο έλεγχος και η εποπτεία έρχονται κάπως καθυστερημένα σε ό,τι φορά τις διαδικασίες της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαφάνεια γιατί η διαφάνεια είναι ταυτόχρονα ένα είδος μηχανισμού ελέγχου από όλους ε, τους φορείς της αγοράς και τη διαφάνεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι καταναλωτές για να ελέγξουν την κατάσταση στην αγορά. Η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση με ένα δημοσιογράφο που είπε ότι αυτό είναι κατά της εσωτερικής αγοράς όταν μιλήσαμε για τη διαφάνεια. Όταν όμως θέλουμε αποτελεσματική αγορά, πότε έχουμε αποτελεσματική αγορά, όταν οι, διάφοροι παράγοντες έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Αυτό ισχύει για τα παράγωγα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το πρόβλημα με τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, προκλήθηκε από την αδιαφάνεια που επικρατούσε. Δεν ήταν εμφανείς αυτές οι συναλλαγές. Ήταν ε, συναλλαγές μεταξύ των ενδιαφερομένων, αλλά δεν ήταν προφανής ο κίνδυνος, δεν ήταν ορατός ο κίνδυνος για τους υπόλοιπους μετόχους στην αγορά όταν κλονίστηκε αυτή η χρηματοπιστωτική πυραμίδα και η διαφάνεια συνέβαλε σε αυτό. Τώρα έχουμε το θέμα του ρόλου των οίκων αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, και μάλιστα δεν υπάρχει καμία προσωπική υπογραφή ε, κάτω από μια ε, γνωμοδότηση και μπορεί να, να ρίξουν και ολόκληρη η κυβέρνηση ή να, να, οδηγήσουν, να καταβαραθρώσουν και ολόκληρη η χώρα. Θα πρέπει να αναλαμβάνετε μια ευθύνη. Εμείς είμαστε υπόλογοι. Έχουμε λογοδοσία, ενώ η πίστη ή και αυτή η πιστοληπτική ικανότητα κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Δεν ξέρουμε ποιο ετοιμάζει την έκθεση και τα αποτελέσματα των εκθέσεων αυτών είναι μερικές φορές ε, ολέθρια. Επίσης, ε, έχουμε, ε, γίνονται μερικές φορές καταθέσεις αν οι προβλέψεις τους επι, ε, αν ε, δίνουν μια εγγύηση σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψει του να την λαμβάνουν, σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν να τι κάνουν. Αν είχαμε κάτι τέτοιο, θα είχαμε μεγαλύτερη ίσω ευθύνη και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με το θέμα της εποπτείας. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει στις δημόσιες συμβάσεις να υπάρχουν ρήτρες ότι ένα τμήμα των δημόσιων συμβάσεων να, να τον αναλαμβάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί να μην έχουμε τέτοια ρήτρα για να προωθήσουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις. Αναφέρθηκε το θέμα των Κινέζων. Ε, Τελικά δεν έγιναν αυτές οι αναθέσεις στους Κινέζους. Οπότε δεν βγήκαν κερδισμένοι οι Κινέζοι από αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ε κυρίου για το ενοχικό δίκαιο, νομίζω ότι η Πολωνική Προεδρία είπε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα δικαιώματα των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και αν λάβει αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβάλει το νομοθετικό σχέδιο, θα ξεκινήσουν οι εργασίες και επίσης αυτά θα τα εξετάσει η Πολωνική Προεδρία, λαμβάνοντα υπόψη και την θέση της Επιτροπής σας, αλλά και τη θέση των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ερωτήσεις της κυρίας Ρουζατούν, θα ήθελα να σας παραπέμψω στο σχέδιο για τον αναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μπορεί να μην είναι τόσο ορατό αυτό το σχέδιο όσο η περιαγωγή, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, ένα πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς. Για παράδειγμα, βλέπουμε μερικές φορές ε, τι προβλήματα έχουν με διασυνοριακές συναλλαγές και τι παράπονα λαμβάνουν οι οργανώσεις καταναλωτών. Δεν υπάρχει δυνατότητα διερεύνηση μερικών υποθέσεων και ικανοποίηση των απαιτήσεων. Αν λύσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα με τον εναλλακτικό μηχανισμό διακανονισμού των διαφορών, θα έχουμε πραγματικά ένα απτό αποτέλεσμα για του πολίτε. Ε, έχουμε άλλα τρία θέματα σήμερα για να συζητήσουμε ε, πριν ε, κλείσουμε τη σημερινή ημερίδα και ξέρω και ότι ο κύριος Αντιπρόεδρος πρέπει να πάει σε μια άλλη συνάντηση. Ελπίζω την επόμενη φορά να μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και θα ήθελα απλά να σας επιδώσω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό το δίνω σε εσά ε, είναι μελέτη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Συζητήσαμε για αυτήν σήμερα το πρωί ε, και σα δίνω και ένα αντίγραφο ε, με το ενημερωτικό δελτίο για την κοινή αγορά. Εκεί είναι και η δική σα προσωπική φωτογραφία. Σα το επιδίδω λοιπόν αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και μα απευθύνετε το λόγο. Uh, um, Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα. Έχουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Στάιλερ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Προγραμμάτων. Και πρέπει να το δούμε για να προετοιμάσουμε τροπολογίες για το Σεπτέμβριο. Ορίστε κυρία Στάιλερ. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Ευχαριστώ όσους συνεχίζουν. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια νέα μέθοδος για την προώθηση του συντονισμού των προγραμμάτων που αφορούν τη δέσμη της οικονομικής διακυβέρνησης. Η συνάδελφος Περβάνς Περέζ είναι αρμόδια συντάκτρια της ε, έκθεσης από την Επιτροπή Οικονομικών. Εγώ θα καταθέσω μερικές δικές μου τροπολογίες, αλλά τα σημαντικότερα έχουν ήδη κατατεθεί. Ήθελα να χρησιμοποιηθούν οι εκθέσεις της δικής μας Επιτροπής και τα εργαλεία όπως το scoreboard της εσωτερικής αγοράς γιατί η Κομισιόν πρέπει να διαβουλεύεται με όλες τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τακτικά. Και αντί να γράφει απλώς μια έκθεση θα έπρεπε να διασφαλίζει ότι ακούγονται όλες οι προτάσεις και συστάσεις. Όπως και οι γνωμοδοτήσεις από τις άλλες επιτροπές μιλάω και εγώ για την κοινωνική συνοχή και στην παράγραφο 6 για αυξημένη προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είπα λοιπόν ότι θα καταθέσω ορισμένες τροπολογίες και θα ήθελα αν θέλουν οι συνάδελφοι να έρθουν σε επαφή με το γραφείο μου αν θέλουν να συμπεριληφθεί κάτι ή αν έχουν απορίες. Είναι πολύ σύντομη γνωμοδότηση. Εξετάζει Ποιο είναι ο ρόλο τη ΣΥΜΚΟ για την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και ελπίζω να τη δέχονται όλες οι ομάδες. Η διορία για την κατάσταση τροπολογιών λήγει στις 20 Ιουλίου και θα εξεταστεί στις 19 Σεπτεμβρίου στην στην 22 Σεπτεμβρίου για να περάσει με τελικά το θέμα στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρθηκαν και που παρέμειναν μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Στάιλερ. Κυρία Γκάλο τώρα η Σκιώδης από το ΕΛΚΟ, κύριος Κρόιτσμαν και είμαι και εγώ Σκιώδης, και εγώ. Η κυρία Γκάλο όμως πρώτη. Α, και ο κύριος Διόνι βέβαια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την εισηγήτριά μας για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που είναι σαφές, περιεκτικό και πλήρες. Οι κρίσεις που ζήσαμε και αυτή που ζούμε ακόμη τώρα έδειξαν ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη συντονισμού των οικονομικών προγραμμάτων. Τον περασμένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τους δύο στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επαλήθευση της εφαρμογής των ε, μέτρων για δημοσιονομική πειθαρχία των χωρών και του προγράμματος 2020. Το έξι σημεία που προτείνει το σχέδιο γνωμοδότης της Κατερίνη Στάιλερ, ε, θα ήθελα να τονίσω δύο προτεραιότητες. Πρώτον, να υποβοηθηθεί η δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τέτοιου είδους ώστε να διασφαλίζει σχέσεις που θέλουμε να έχουμε όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες και την Κίνα. Πρέπει δηλαδή να εφαρμοστούν ρήτρες αμοιβαιότητας με τις τρίτες αυτές χώρες, αυτό μου φαίνεται προφανές και σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της φορολογίας παραδείγματο χάρη τους, ε, τα ποσοστά του ΦΠΑ που τελικά συνιστούν άνηση μεταχείριση για τα ψηφιακά αγαθά. Άλλο σημείο που μου φαίνεται επίσης ζωτικό στη γνωμοδότηση αυτή είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διότι ξέρουμε ότι εκπροσωπούν το 90% του επιχειρηματικού ιστού και θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα να καταπολεμηθούν οι απομιμήσεις, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι διαμεθοριακές πληρωμές, να μειωθούν τα διοικητικά άχθη και να αναπτυχθούν δίκτυα ενεργειακά και άλλα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ συμφωνώ με την ε, συντάκτρια της ε, εισήγησης ότι πράγματι η κοινή αγορά πρέπει να αντιλαμβανθεί σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ε, καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχουν αυτοί οι βασικοί στόχοι για το 2011 και το 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα επιληφθεί και αξιολόγησε την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη σε έξι από τα προτινόμενα μέτρα για την επίτευξη του στόχου. Πρόκειται όμως για δηλώσεις προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση και οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη δεν παίζουν πια κανένα ρόλο. Η Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη για το θέμα της ε, κοινή αγοράς και παραθέτω περαιτέρω στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, κυρίως ε, με την άρση των εμποδίων στις, ε, στα ελεύθερα επαγγέλματα και στις ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές. Αυτό που προκύπτει είναι λίγο φτωχό. Η ανακοίνηση Κομισιόν για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιορίζεται κυρίως ε, σε αυτά τα θέματα, ενώ υπάρχουν και άλλα δύο, όπως καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις και περιορισμός της γραφειοκρατίας σε δημόσια συμβάσεις. Επειδή δεν έχουμε χρόνο θα περιστώ σε ένα και μόνο θέμα. Ε, υπάρχει ένα θέμα στην ημικό που δεν το παίρνουμε πολύ σοβαρά, όμω δεν το βρίσκω σωστό ε, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, δυστυχώς αυτό αναφέρεται και στην έκθεση, ε, να λέμε ότι για όλα ε, πρέπει να γίνουν εισηγεί. Παίρνω με το θέμα τη Ελλάδα. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε στους Έλληνες πρέπει να κάνετε οικονομία, να καλύπτετε τις προποθέσει και από την άλλη η Κομισιόν να μην λέει τι κάνει εκείνη για να βοηθήσει τους Έλληνες να προχωρήσουν. Δηλαδή, όταν ε, δεν υπάρχει πρόγραμμα ανάκαμψης, όταν η Επιτροπή ε, δεν ε, λέει ότι δεν επιθυμούμε τη συγχρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα. Να λέμε μόνο ευρωπαϊκό εξάμεινο και να βλέπουμε μετά κατά πόσον αυτά τα οποία ελέγχθησαν τηρήθηκαν ή όχι, αλλά το να μην λέει να μην αναφέρεται ποιο, ποια είναι η συμβολή της Κομισιόν για να βοηθήσει το πλαίσιο υποτίθεται της πολιτικής συνοχής, αυτό το βρίσκουμε πολύ φτωχό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήταν σωστό ε, στις, ε, στην έκθεση αυτή να μην λέμε μόνο ότι η Κομισιόν είναι αναγκασμένη να υποβάλει προτάσεις, αλλά να, εκθέσεις, αλλά να υποβάλει και προτάσεις για το ε, πώς ακριβώς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν αυτά που λέγονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, εξοικονόμηση, αποταμίευση, αποταμίευση, ε, μείωση ε, χρέους, γιατί το να επιβάλλουμε μόνο περιορισμού στα κράτη-μέλη αυτό δεν βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήμασταν ευγνώμονες εάν στη γνωμοδότηση μπορούσατε να συμπεριλάβετε κάτι σαν και αυτό που σας είπα τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα καταθέσετε σχετική τροπολογία, λέει ο πρόεδρο, Και εκ μέρου τη ομάδα μου να σας πω ότι η κυρία Στάιλερ έκανε ακριβώς αυτό που θέλουμε να κάνει η Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι η Πολωνική Προεδρία είπε υπό τη δική τους την Προεδρία θα ελέγχουν τις 12 ε, δράσεις ε, και αυτό ε, πρέπει να ε, αναφερθεί. Το άλλο το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε είναι ε, το βαθμολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί κοιτάζοντας λιγάκι στοιχεία που αφορούν στον ανταγωνισμό και στα ωφέλη από τον ανταγωνισμό αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι και γι' αυτό λοιπόν ε, και αυτό μπορείτε να το συμπεριλάβετε. Νομίζω λοιπόν ότι η συνεισφορά σας ήταν πολύ σημαντική ε, και θεωρώ ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόεδρο. Ε, ο κύριος Διγιόν, ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Εγώ μπορώ να είμαι πολύ σύντομος διότι μόλις είπατε αυτά που θα έλεγα κι εγώ. Δηλαδή ότι υπάρχει και το θέμα της πληροφόρησης των καταναλωτών. Η ομάδα μου ενδιαφέρεται για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά η έκθεση αυτή μας ικανοποιεί. Όλοι συμφωνούμε δηλαδή ότι είναι απαραίτητο να συνδιαχειριστούμε και την ενιαία αγορά. Επομένως, οι προτάσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν και την ίδια την Κομισιόν για να βελτιώσει την πρόταση της. Ο εισηγητής έχει τη στήριξή μου, τον ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλά, δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Αναμέναμε τον κύριο Σούλτς από την Κομισιόν, δεν ήρθε. Θα μας μιλήσει άλλη φορά. Νομίζω όμως ότι είχαμε πληροφορήσει την Κομισιόν. Τέλος πάντων, κυρία Στάιλερ θέλετε να καταλήξετε γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε στο αεροδρόμιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους Κιώδης για αυτή την αρχική ανταλλαγή απόψεων και για τις τροπολογίες τους που αναμένω. Βέβαια χρειάστηκε να περιοριστούμε στους τομείς όπου έχουμε δικαιοδοσία στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό uh, Γι' αυτό νομίζω ότι όλες οι προτάσεις που έγιναν θα γίνουν δεκτές, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη η πίεση χρόνου, οι σημερινές συστάσεις νομίζω ότι ενδυναμώνουν το δικό μου κείμενο. Μπορεί να διαφωνώ με την κυρία Γκάλο αν για μία και ένα κοινό ποσοστό ΦΠΑ αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή μας και η δουλειά που κάνουμε εδώ θα διασφαλίσουμε να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και αυτό νομίζω οι πολίτες το θέλουν. Πολύ ωραία. Στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε, το είπατε κι εσείς. Ωραία. Και τώρα άλλο τεράστιο θέμα για τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα. Κύριε Βαντεκάμπ, είστε εκεί πίσω. Ελάτε πιο μπροστά. Ελάτε πιο μπροστά. Καθίστε μπροστά για να σας βλέπουμε πιο καλά. Είναι οι είναι. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Εγώ είμαι εδώ, ο Ραβίνη λείπει. Ο κύριος Γκίλαν, να δεν από τη Γενική Διεύθυνση των Επιχειρήσεων. Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Ματίνο λείπει, τι να κάνουμε. Ορίστε κύριε Βαντεκάμπ μου. Έχουμε βλέπω 300 τροπολογίες. Μίλησα με τον Κώστα. Πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση σήμερα, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος και για δεύτερη, δεύτερο κύκλο συζητήσεων μετά τα διακοπάς. Σήμερα λοιπόν θα είναι απλώς η πρώτη φάση, οι πρώτες σας απαντήσεις των σχολείων από τους Σκιώδης. Και θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε περισσότερη ώρα μετά τον Αύγουστο. Γιατί πρέπει να δούμε και με το Συμβούλιο τι θα γίνει. Μήπως απλώς να μας ενημερώσετε για τις τελευταίες εξελίξεις. Ορίστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τους ε, Σκιώδης, αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους που κατέθεσαν ε, τροπολογίες. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που κατατέθηκαν τόσες πολλές ε, τροπολογίες γιατί τελικά τι γίνεται, πιστεύει κανείς ότι έχει κάνει μια πολύ καλή έκθεση ε, και ξαφνικά ε, κατατίθεται ολόκληρη πλημμυρίδα τρομολογιών. Τέλος πάντων, ε, αυτό βέβαια από την άλλη υποδεικνύει ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ ως Επιτροπή για την έκθεσή μου. Και εγώ το καλοκαίρι μου όλες μου τις διακοπές θα τις περάσω προσπαθώντας να εξετάσω αυτές τις τροπολογίες και κάτω από φιλοσοφικό πρίσμα. Τέλος πάντων, Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε και αύριο ακόμα. Γιατί αν συγκρίνει κανείς τις τροπολογίες ανάμεσά του θα δει ότι η μία ακυρώνει την άλλη. Από τη μια υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να προχωρήσουμε γρηγορότερα, από την άλλη εκείνοι που επιθυμούν ε, να καθυστερήσουμε λιγάκι. Αλλά όπως ξέρετε εγώ είμαι ε, Πραγματικό ακρεφνής δημοκράτη, και γι' αυτό λοιπόν το καλοκαίρι σας είπα θα πάρω τι τροπολογίες, θα τι μελετήσω και ελπίζω ε, να μπορώ να συνεργαστώ και με τους σκιώδεις εισηγητέ. Τι ε, τροπολογίες ε, τις έχω ομαδοποιήσει και καλύπτω βασικά 10 τομεί. Θα τα πω σύντομα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Το σημαντικότερο είναι οι εκπομπές ε, και τα χρονοδιαγράμματα που πάνε με τις ε, εκπομπές του. Η δεύτερη ομάδα ε, των τροπολογιών αφορούν τα σκούτερ και τα μοτοποδήλατα. Κατόπιν, ο το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος που χρειάζεται για να τοποθετηθούν συστήματα πέδησης στην ε, κατηγορία υπαρθμών 4 είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, η σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και τα κιλοβάτ. Ε, υπάρχουν ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά, ε, τα οποία είναι υψηλής απόδοσης. Αυτό όμως δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας και πρέπει να το δούμε λιγάκι προσεκτικά το θέμα, να εξελιχθεί ο τομέα Η πέμπτη ομάδα είναι τα μέτρα κατά, τις, ε, κατά των παρεμβάσεων τροποποίησης των οχημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, υπάρχει ένας άλλος ε, τομέας και αυτός είναι σημαντικός, οι πληροφορίες για τη συντήρηση. Αφορούν το άρθρο 60 του προτινόμενου διαγωνισμού. Έβδομο, είναι τα τεστ αντοχής ε, που ε, και εσείς ε, τα αναφέρετε. Το περίφημο τεστ Καλιφόρνια και κατόπιν η 8η ομάδα είναι η έγκριση μικρών σειρών οχημάτων. Η κυρία Κόμη έχει μία τροπολογία που αφορά στο βάρος κάποιων ε, κατηγοριών οχημάτων. Η Πιάτζο, ε, παραδείγματο χάρη, ε, προσπαθεί να αυξήσει το βάρος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και τέλος πρέπει να στήσουμε την τροπολογία του κύριου Μάντερς, την 238, που αφορά στους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους. Αυτές είναι οι 10 ομάδες τροπολογιών όπως ε, τις έχω μοδοποιήσει εγώ τις ε, τροπολογίες. Πρέπει να βρούμε λοιπόν συμβαστική πρόταση για αυτές ε, τις τροπολογίες κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Θέλω να κάνω και μία παρατήρηση για το Συμβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία που με βοήθησε να καταθέσω την πρόταση. Και δεύτερον, εύχομαι στην Πολωνική Προεδρία καλή επιτυχία στις προσπάθειές της να προχωρήσει περαιτέρω την πρόταση. Εξ όσων γνωρίζω, η Ουγγρική Προεδρία και οι Ουγγρικές προσπάθειες είναι εκείνες που βοήθησαν στο να επιληθούν πολλά προβλήματα και να μπορεί να προχωρήσει η πολιτική προεδρία. Um, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπορείτε να έχετε χρόνο για να μελετήσετε, αλλά θα μπορείτε σίγουρα να έχετε χρόνο για να συντάξετε ε, πάρα πολλές αλλαγές. Ας ε, δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ε, σκιώδεις για να τοποθετηθούν σε αυτές τις ομάδες τροπολογιών σύντομα και χαιρετίζουμε αυτά που είπατε ότι επιθυμείτε τον συμβιβασμό. Θα βρούμε λοιπόν ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, ίσως τον Αύγουστο, να μπορείτε να καταθέσετε τις συμβαστικές προτάσεις ε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για το θέμα και μας ε, παρακολουθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καπ και έτσι κανείς ε, μπορεί να περάσει το καλοκαίρι του. Αντί να τρέχει με τη μοτοσυκλέτα του, να ασχολείται με τροπολογίες για μοτοσυκλέτες. Καλή και αυτή η εναλλακτική λύση. Εγώ δεν θέλω να πω και πάρα πολλά. Το πρώτο θέλω να ευχαριστήσω για την ε, καλή αγαστή συνεργασία που έχουμε εδώ και έξι περίπου μήνες. Εν τω μεταξύ γνωριστήκαμε και πάρα πολύ καλά και θέλω να πω μερικά πράγματα για τις ε, τροπολογίες. Ούτε καν που το πίστευα ότι θα είμαι σε θέση να το πω, θα το πω. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το άρθρο 18 αφορά στα μέτρα για αλλαγές στα οχήματα αυτή την ε, τροπολογία ε, να διαγράψουμε εκεί τις κατεξοδότηση πράξη έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να λάβει τις δικές του τις ρυθμίσεις. Φαντάζομαι δεν θα σας ε, εκπλήξει το ότι ο παράγων ασφάλεια είναι πολύ σημαντικός ε, για μένα και εκεί μπορώ να γίνω μέχρι και ενοχλητική. Ε, το θέμα της πέδησης, ABS, όπως σας έχω πει επανειλημμένα, πράγματι εκεί θα καταθέσουμε τροπολογίες ή τις έχουμε ήδη καταθέσει απεμπλοκή, υποχρεωτική για όλες τις μοτοσυκλέτες από το 2015. Κατόπιν τούτου τα οχήματα ε, τα οποία όμως είναι ε, χαμηλής απόδοσης θα πρέπει να εξαιρούνται. Και εγώ για άλλη μια φορά λέω ότι με τη βοήθεια τεχνολογιών πέδησης μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των ατυχημάτων ε, στις μοτοσυκλέτες και να το περιορίσουμε δραστικά. Ελπίζω και να είμαι και πεπισμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι ότι εντωμεταξύ θα έχετε κι εσείς διαπιστώσει ότι ούτε το υλικό ούτε το κόστος εφαρμογής ε, των συστημάτων πέδησης ε, είναι υπερβολικό, ούτε και ότι αυτά ε, οδηγούν σε μείωση της απόδοσης. Με άλλα λόγια, κάθε θάνατος, κάθε θανατηφόρο ατύχημα από μοτοσυκλέτα μας υποχρώνει να λάβουμε μέτρα. Το σύστημα ABS είναι εκείνο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Κατά τα άλλα προτείνω ε, την κατηγορία Euro 4 και την ε, Euro 5 να τη συνδέσουμε από το 2015 να είναι υποχρεωτική η Euro 4 για, όλες, ε, τους, για όλους τους τύπους οχημάτων. Λιγάκι επιφυλακτική είμαι στη συζήτηση για τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία πρέπει να εξαιρούνται από την έγκριση τύπου. Ε, δεν το βρίσκω αυτό απόλυτα σωστό. Εμείς χαιρετίζουμε το ότι η Επιτροπή προτείνει την έγκριση μικρών σειρών. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι θετικό που πρέπει να το ε, υιοθετήσουμε. Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή ε, συνεργασία. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Βαντερκάμπ, για την πρώτη αυτή έκθεσή του και τον ε, κατέπληξε ο μεγάλος αριθμός τροπολογιών, αλλά αυτή είναι η Ευρώπη. Παλιά ήταν μέλος της ε, Ολλανδικής Βουλής, ε, παρήγαγε νομοθεσία για 15 εκατομμύρια πολίτες, τώρα ασχολείται με νομοθετικά πακέτα που θα επηρεάσουν τη ζωή 500 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο να προσαρμοστεί κανεί. Το σημαντικό εδώ είναι να είναι καλό το αποτέλεσμα. Πάντω η αρχή έχει γίνει και είναι θετική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. γιατί μπορεί στην αρχή να υπήρχε ένα πρόβλημα τη τροπολογίες παρά την ε, καθυστέρηση και χάρη στι προσπάθειε της γραμματείας ε, ρυθμίστηκε το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τα μοτοποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην Κίνα και έχουμε πολλά ατυχήματα με αυτά τα ηλεκτρικά οχήματα γιατί είναι και σχεδόν αθόρυβα αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα και μάλιστα αυτά τα πολύ ελαφρά οχήματα, τα ηλεκτρικά, ε, σκέφτονται να τα απαγορεύσουν και στην Κίνα εξαιτία του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων. Το θέμα είναι να είναι και ασφαλίστερα τα οχήματα. Είναι ένα από τα μελήματα αυτής της πρότασης και δεν ξέρω ποια θα είναι η περιοδικότητα που θα επιλέξουμε, δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Πάντως θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνεται ένας έλεγχος και ένας αναγνωρισμένος ε, ε, τεχνικός να προβαίνει στον τεχνικό έλεγχο για να εξασφαλίζεται η σωστή κατάσταση, η επισκευή του οχήματος. Θα υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες ώστε να γίνει ευκολότερη η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Μιλήσαμε για το σύστημα πέντησης ABS και καλό θα να προσθέσουμε και άλλες καλύτερες πρακτικές, γιατί σήμερα το ABS είναι η καλύτερη τεχνική ρύθμιση, αλλά στο μέλλον μπορεί να έχουμε ακόμη πιο προηγμένες τεχνολογίες. Επίσης αναφέρεται υποχρέωση πληροφόρησης των παραγωγών. Θα πρέπει να είναι λογική αυτή η υποχρέωση και το θέμα της αποζημίωσης της αμοιβή. Επίσης θα πρέπει να δούμε και το θέμα των φορτίων, να μην, να μην υπερβάλλουμε και σε αυτό. Πάντως ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και θα καταλήξουμε σε αίσιο αποτέλεσμα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί και η πλευρική ορατότητα, γιατί πολύ συχνά η τα ατυχήματα με μοτοσυκλέτες ε, οφείλεται στο γεγονό ότι δεν τους βλέπουν οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι εδώ η κυρία Ρούλα, οπότε θα σχολιάσω εγώ. Έτσι λίγο το ιστορικό. Καταρχήν, έχουμε προτείνει στον εισηγητή να χειριστεί το θέμα των τετρακίνητων αυτοκινήτων των... γιατί ο μεγάλος αριθμός τους χρησιμοποιείται για πολύ συγκεκριμένη χρήση αυτό σχετίζεται και με την έκθεση Παντσέρη χρησιμοποιούνται περισσότερο από γεωργούς Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα θεωρήσουμε ως γεωργικάς μηχανάς. Από την άλλη υπάρχει ένα πρόβλημα διαφοροποίησης του κάθε τύπου. Ένα επαγγελματικό δασοκομικό όχημα πώς διαχωρίζεται από ένα επαγγελματικό γεωργικό καμιά φορά είναι τα ίδια. αλλά η διαφοροποίηση θα μπορούσε να επιτρέψει σε ορισμένα από αυτά να χρησιμοποιούνται και στις δημόσιους δρόμους. Ενώ τα οχήματα που κυκλοφορούν μόνο σε δασικά μονοπάτια δεν έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν στον δημόσιο δρόμο. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας το λύσει. Έπειτα δόθηκε μεγάλη προσοχή σε μερικά συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα ώστε οι κανονισμοί να είναι πιο αποτελεσματικοί αλλά και να μειωθεί το κόστος της εφαρμογής τους χωρίς να μειωθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η Κομισιόν μερικές φορές ακολούθησε το παράδειγμα βαρεωτέρων οχημάτων ενώ τα ελαφρότερα όπως τα μοτοσακό ας πούμε τα σκούτερ δεν μπορεί να έχουν την ίδιες διατάξεις. Πρέπει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί μειώνεται η αποτελεσματικότητα των οχημάτων ως προς τις εκπομπές διοξιδίου. Στην Αμερική έχουν καθορίσει ορισμένα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά τον μηχανικό έλεγχο του αυτοκινήτου και εφαρμόζουν έναν παράγοντα, ένα πολλαπλασιαστή. Έτσι θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σωστά τον ισχύοντα κανονισμό αφού πρώτα καθοριστούν δηλαδή τα σωστά πρότυπα. Μου φαίνεται λογικό το αμερικανικό παράδειγμα γιατί αν εφαρμόσουμε αυτούς τους συντελεστές μείωσης της αποτελεσματικότητας μπορεί τελικά να μειωθεί και το κόστος κατασκευής των οχημάτων αυτών. Μετά η διαγνώση, τα έλεγχη αυτό είναι κάτι γενικότερο που θα ήθελα να το συμπεριλάβει ο εισηγητής. Δεν υπάρχει καμία πραγματική εξήγηση κόστους ωφέλους για αυτά που θέλει να εφαρμόσει η Κομισιόν. Ένα από αυτά τα προβλήματα, το οποίο βέβαια είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα δεν πρόκειται να είναι το μόνο, είναι ότι για τις διαγνώσεις που γίνονται από το ίδιο το αυτοκίνητο στον πίνακά του πρέπει να εμφαίνεται και ο τρόπος εκπομπής των καυσαερίων. Η περιβαλλοντολογική επίπτωση δεν είναι σχετική εδώ, γιατί εδώ μιλάμε για τα ελαφρότερα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι θα κόστιζε 9 εκατομμύρια για να επιτευχθεί όφελος ενός εκατομμύριου. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, το λέω και στην κυρία Βέστφαλ. Δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι το ADS είναι αποτελεσματικό και για τα μοτοσακά. Πιστεύω ότι το combined braking system είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η πρόταση που το αφορά για τα σκούτερ λειτουργεί συνεχώς. Όχι μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις, αλλά και στην κανονική του χρήση. Και αυτό είναι πολύ πιο ωφέλιμο. Πρέπει εδώ να ακούσουμε εμπειρογνώμονες. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα το άλλο σύστημα είναι καλύτερο. Χρειάζεται εδώ μια τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Και τότε αν υπάρξει αυτή μπορεί να πιστέψω, να πιστώ. Αυτά είναι τα κυριότερα σχόλια που ήθελα να κάνω. Υπάρχουν βέβαια και άλλες λεπτομέρειες αλλαγές, αλλά ελπίζω ο κύριος Βαντεκάμπ να πιστεί ότι αυτά τα σχόλια οφείλονται στο ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά την έκθεσή του. Κανείς άλλος, καμία άλλη. Η Κομισιόν. Ξέρω ότι και εσείς έχετε πάρει μέρος στη συνεννοήση με τον κύριο Βαντενκάμπ. Μήπως θέλετε να κάνετε κανένα σύντομο σχόλιο. Αλλιώς μπορούμε άλλη φορά να σας ακούσουμε. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον κύριο Ρέντες που αντικαθιστά τον κύριο Ματίνο. Συντομότατα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να τις ταξινομήσουμε σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, ενδιαφέροντων. Εκτός από τους δέκα λοιπόν αυτούς τομείς που ταύτισε και ο εισηγητής που αφορούν σαφώς την πρότασή μας. Υπάρχουν και μερικές που ξεπερνούν κατά πολύ το εύρος και το στόχο της οδηγίας. Και πρέπει να προσέξουμε να μην βγούμε εκτός θέματος και λύσουμε να, να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της πρότασης και σε άλλα οχήματα. Επίσης, Ήδη ανησυχούμε για μερικές τροπολογίες που ζητούν μείωση ή περιορισμό των περιβαλλοντολογικών προτύπων που θέλουμε να εφαρμοστούν. Αυτό θέλουμε να, να συζητηθεί και να υπάρξει νέα συνεννόηση με τον εισηγητή ώστε να βρεθεί καταλληλότερη λύση και φυσικά όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Βαντενκάμπ θέλει ακόμη πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή αξιολόγηση όλων των τροπολογιών και περιμένουμε τις συμβιβαστικές που θα μας ετοιμάσει για μετά τις διακοπές ο κύριος Βαντενκάμπ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαντενκάμπ. Θέλετε να καταλήξετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει εδώ ένα πεδίο μάχης ή μάλλον καλύτερα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα παρακολουθήσω τη συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και τη κυρία Βέσφαλ και θα δούμε αν μπορούμε να συντάξουμε μια συμβαστική πρόταση. Πάντως νομίζω ότι τα θέματα είναι σαφώς προσδιορισμένα, διευκρινισμένα και είναι όλα φυσικά σοβαρά. Θα πρέπει να δούμε πότε θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας παρατήρηση, όντως είναι περίπλοκο το πρόβλημα και υπάρχουν ε, ε, κάποια οχήματα που ε, ναι ε, είναι προορισμένα για την γεωργία, αλλά τα χρησιμοποιούν και στους, στους δρόμους, στα περίφημα quad, τις γουρούνες, που κανονικά δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους, γιατί είναι επικίνδυνα οχήματα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ του σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, αυτά τα quad, αυτές οι γουρούνες, δεν θα πρέπει να περάσουν ε, στην τυποποίηση των μοτοσυκλετών Πάντως και με τη δική σας βοηθό θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ικανοποιητική για όλους συμβαστική λύση. Σας ε, εύχομαι καλό καλοκαίρι και ό,τι όχημα και χρησιμοποιήσετε δίτροχο, τρίτροχο ή τετράτροχο, προσοχή στο δρόμο. Καλώς θα επανέλθουμε στην εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών. φυσικά τα εκπροσωπώ τους και οδησηγητές ότι σας ευχαρίστησα για την ανοιχτή σας προσέγγιση, το συνεργάσιμο πνεύμα σας και το, τη διαλλακτικότητά σας. Και περιμένουμε να συνεργαστούμε στις συμβαστικές λύσεις. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση κυρία Ιβάνοβα. Αφορά το μέλλον του ΦΠΑ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Έχουμε εδώ και γιατί τον κύριο Κορέα Δεκάμπος. Φαντάζομαι ότι ο ακαταπώνητος ε, κύριος Κρόιτσμαν αντικαθιστά τον κύριο Μπουσόη. Δεν έχουμε πράσινο. Ο κύριος Διόν είναι παρόν. Κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, ο κύριος Νίλ. Παρίσταται υπάρχει εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης για τη φορολογία. Α, ο κύριος Ραπώνη, ο κύριος Ραπώνη εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας. Καλώς ήρθατε. 12 λεπτά μας έχουν απομείνει. Θα προσπαθήσουμε να σας τριμώξουμε και εσάς εκεί πέρα. Η κυρία Ιβάνοβα. Ελπίζα να έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά λακωνική. Είναι σαφέστατο ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε τεράστιες προκλήσεις για τα οικονομικά των κρατών μελών. Πολλέ χώρες αύξησαν του συντελεστέ ΦΠΑ ή σκέφτονται να του αυξήσουν αισθητά, είτε ω αντίδραση στην κρίση, είτε στο πλαίσιο μια πιο μακροπρόθεσμες αλλαγή στην φορολογική του στρατηγική. Η γνωμοδότησή μου επικεντρώθηκε σε πολλά και διάφορα θέματα. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω τέσσερα από αυτά μόνο. Το πρώτο αφορά την ε, περιπλοκότητα των ε, ισχυουσών διατάξεων για το ΦΠΑ και τα διοικητικά εμπόδια. Γι' αυτό οι επιχειρήσει θεωρούν το σύστημα ΦΠΑ ω εμπόδιο στην ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Ισχύουσε ρυθμίσει για τι ενδοκινοτικέ συναλλαγέ ε, επηρεάζουν αρνητικά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και σίγουρα χρειαζόμαστε κάποια μέτρα για να τις ανακουφίσουμε, να ανακουφίσουμε το βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε πιο αποφασιστικές ε, αλλά και πιο απλές διαδικασίες που θα ε, είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Άλλο φλέγον ζήτημα ε, στην εποχή του διαδικτύου είναι οι διαφορετικέ συντελεστές ΦΠΑ και οι διοικητικές διαδικασίες που δημιουργούν προβλήματα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και για τους Ευρωπαίους λιανοπολιτές κάνουν τη ζωή σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα πώλησης ε, διαφόρων υπηρεσιών. Θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξασφαλίζοντας καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών, μια καλύτερη ε, διαλειτουργικότητα στο θέμα αυτό. Γίνονται συζητήσει πίσω μου και να ε, επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ. Νομίζω ότι έτσι θα διευκολυνθούν οι διασυνοριακέ διαδικασίε ΦΠΑ και έτσι θα διευκολυνθούν πρώτα απ' όλα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Τέλο, ε, θα επισημάνω κάτι που κατά τη γνώμη είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας σε οποιαδήποτε απόφαση για μειωμένου συντελεστέ ΦΠΑ. Τετοιε αποφάσει θα πρέπει να επαφείται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη να διαφυλάξουν την κυριαρχία τους ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για μειωμένου συντελεστέ σε ορισμένου τομεί, προκειμένου να εφαρμόσουν καλύτερα τι κοινωτικές και εθνικέ πολιτικέ με βάση του διαφορετικού εθνικού, ιστορικού οικονομικού, κοινωνικού ή περιβαλλοντικού λόγου. Mm και παράγοντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κοιόδης συγκητές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση που είχαμε στο Στρασβούργο, που πραγματικά ήταν ικανοποιητική και επικοδομητική και περιμένω και πάλι τα σχόλιά τους και δεχομένω και κάποιες συμπληρωματικέ προτάσεις για την γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Ε, λυπάμαι που δεν μπορώ να σα διαθέσω 20 λεπτά, αλλά καλύψετε το θέμα πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ο κύριο Κορέντε Κάμπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συνάδελφο κυρία Ιβάνοβα και να την ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας έδωσε στο Στρασβούργο να συζητήσουμε με τους σκιώδεις ηγητές το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ελάχιστα είναι τα σχόλιά μου, κάποια συμπληρώματα περισσότερο. Όντως, ο ΦΠΑ ε, πέρασε, ε, αντικατοπτρίζει την τάση μετάβασης από την άμεση φορολογία στην άμεση φορολογία και έγινε και το βασικό εργαλείο διόρθωση των μακροοικονομικών πολιτικών. Αυτό το νέο χαρακτηριστικό που απέκτησε ο ΦΠΑ με την αύξηση μείωση των συντελεστών και τη σημασία που απέκτησε ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να επισημαθεί στην έκθεση. Κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό είναι η σύγκληση μεταξύ του online περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος, ε, του πραγματικού περιβάλλοντος. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ό,τι αφορά τη συζήτηση για τους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ. Ε, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι είναι σημαντικό να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας και να αφήσουμε την εθνική κυριαρχία για τη λήψη των αποφάσεων αλλά να μην ξεχάσουμε και την ανάγκη να έχουμε κάποιες ε, ενιαίες πλατφόρμες ε, για το ΦΠΑ και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ζητήσουμε μία τυποποίηση του ευρωπαϊκού τιμολογίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, ίσως θα μπορούσαμε εδώ, ε, μια και πρόσφατη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για την, για την περίοδο του 2014-2020 δημιουργία φορολογικού ΦΠΑ για να ενισχυθούν τα κοινοτικά έσοδα, να κάνουμε μια μνή αυτή τη πρόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο δημοσιονομικό πολιτέ πλαίσιο να αναφερθεί και αυτή η πρόταση για την θέσπιση ενό ευρωπαϊκού ΦΠΑ. Ευχαριστώ κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και Θέλω να προσθέσω ότι το ΦΠΑ έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην κοινή αγορά. Ένα αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ μπορεί να συμβάλλει στην εμβάθυνση της κοινή αγοράς. Ε, το κόστος που προκύπτει από το ΦΠΑ και κυρίως από την απόδοση του ΦΠΑ ε, είναι ένα εμπόδιο για την κοινή αγορά. Η Κομισιόν έχει καταθέσει ορισμένες εναλλακτικές λύσεις για ένα μόνιμο σύστημα ΦΠΑ. Ε, βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα αποφασίσουν. Η Επιτροπή αυτή πρέπει να επιμείνει στο ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα όταν είναι το σύστημα απλό και να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να συλλέγουν το ΦΠΑ αποτελεσματικά ε, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες ε, ε, πράξεις ε, με ισοτιμία. Το θέμα της επικουρικότητας είναι πολύ σημαντικό, όμως τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες συντονισμού, κυρίως για τις εξαιρέσεις, απαλλαγές από ΦΠΑ. Αυτό θα διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές. Επίσης, ο Κρίστιαν θέλει να αναφερθεί σε μειωμένο ΦΠΑ για πολιτιστικά αγαθά Υπάρχει ασυνέπεια όσον αφορά την αντιμετώπιση του ΦΠΑ ε, όσον, όταν πρόκειται για ένα αντικείμενο που πουλιέται online, εκεί ισχύει το κανονικό ΦΠΑ, αλλιώς όχι. Αλλά θα πρέπει όμως ε, να προσαρμοστεί η αντιμετώπιση προϊόντων online και offline με τον ίδιο τρόπο. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλούστερο σύστημα ΦΠΑ που σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη μείωση του περιτού γραφειοκρατικού άχθους. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο αν πραγματικά επιθυμούμε διασυνοριακές συναλλαγές ε, να γίνουν αυτές ε, πιο αποτελεσματικές. Η τυποποίηση των υποχρώσεων ΦΠΑ είναι επίσης ευκταία. Βεβαίως πρέπει να έχουμε κατά νου την επικουρικότητα. Ο Κρίστιαν υπέρ του να υπάρχει μια στάνταρ δήλωση ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά γνωρίζει βέβαια ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να το δεχτούν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό τάσεται υπέρ του να υπάρχει ένας εξαντλητικός ε, κατάλογος υποχρεώσεων ΦΠΑ. Και με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ε, θα γνωρίζουν ε, τι τις περιμένει και θα διευκολυνθεί η συλλογή ΦΠΑ. Και ένα άλλο θέμα που θέλει να δείξει ο Κρίστιαν είναι τα νομικά εργαλεία. Μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει την οδηγία για να αφήσουμε κάποιο περιθώριο στα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτό οδηγεί σε ασυνέπειες πλευράς κρατών μελών ε, στην ερμηνεία και αυτό μπορεί να στρεβλώσει την κοινή αγορά. Γι' αυτό είμαστε περισσότερο υπέρ ε, ενός κανονισμού και όχι τόσο οδηγία, γιατί με τον τρόπο αυτό θα επικρατήσει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις επιχειρήσεις. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντιγιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σχόλια. Πρώτον, ένα πρακτικό πρόβλημα Συνήθως λέμε ότι καλό είναι οι άμεση φόροι να γίνουν έμεση γιατί συλλέγονται ευκολότερα. Αυτό δεν το βλέπω όμως στη γνωμοδότηση. Υπάρχει μια γνωμοδότηση γι' αυτό της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχουν απάτες με τον ΦΠΑ και ότι αυτό αφορά και την εσωτερική αγορά. Η ομάδα μου ξέρει πολύ καλά η συνείδηση του γεγονότος ότι οι έμεση φόροι αφορούν, χτυπάνε, ζημιώνουν κυρίως τους φτωχότερους. Για την πρώτη λοιπόν παράγραφο εμείς έχουμε δυσκολία και θα κάνουμε σχετικό τροπολογία. Μάλιστα. Η κυρία Ιβάνοβα συγκέντρωσε απλώς την προσοχή της στα θέματα που ενδιέφεραν περισσότερο τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Οι προτάσεις της για το ΦΠΑ εκεί μέσα εγγράφονται. Επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Κρόιτσμαν για τα προβλήματα που υπάρχουν και τις ανισότητες μεταξύ φορολόγησης των ψηφιακών και των υπολείπων προϊόντων, ιδιαίτερα των ψηφιακών βιβλίων. Γιατί να πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ από ότι τα τυπωμένα. Κυρία Γκάλογα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς για το ίδιο θέμα που δεν το λέει το κείμενο αυτό ήθελα να προσέξει ο εισηγητής και να του πω ότι θα καταθέσω και τροπολογία διότι αν βασιστούμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα ενός ψηφιακού βιβλίου εφόσον ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ως χορήγηση υπηρεσιών φορολογείται με το, στο κανονικό ύψος του ΦΠΑ ενώ το τυπωμένο βιβλίο έχει χαμηλότερο ποσοστό. Και αυτό είχα πει προηγουμένως και στην κυρία Στάιλερ που νόμισε ότι ήθελα ομοιόμορφη ΦΠΑ για όλα και παντού. Όχι. Είναι άνηση μεταχείριση αυτά τα διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ μεταξύ τύπων βιβλίων. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα στο ίντερνετ. Η Κομισιόν λέει ότι θα το σκεφτεί μετά την πράσινη βίβλο της, αλλά εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε το 2015 για να ακουστεί αυτή η λύση, γιατί αυτό προτείνεται θεωρητικά. Νομίζω όμως ότι είναι ουσιώδες να βρεθεί μια λύση πολύ γρηγορότερα. Σας ευχαριστώ που μπόρεσα επιτέλους να μιλήσω. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Κανείς άλλος, καμία άλλη. Να μας πει κάτι η Κομισιόν θέλει, θέλει ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ καταρχήν την κυρία εισηγήτρια για το σχέδιο γνωμοδότησής της που επαναλαμβάνει βασικά αυτά που έλεγε η Πράσινη Βίβλος, η οποία άρχισε μια ολόκληρη συζήτηση. Έχουμε πολλές συμβολές, 1500 ανταποκρίσεις, 8.000 σελίδες. Αναλύουμε, τις αναλύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δείχνει σαφώς ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εσωτερική αγορά. Για το ΦΠΑ η διάσταση της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική γιατί η εσωτερική αγορά είναι το νομικό υπόβαθρο της προόδου του ΦΠΑ. Για συγκεκριμένα θέματα τώρα όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία βεβαίως θα ακούσουμε, θα επαληθεύσουμε ό,τι ακουστεί γι' αυτό και η Κομισιόν θα λάβει τα δέοντα μέτρα και μάλιστα εν καιρό το δέοντι. Αλλά το σύστημα του ΦΠΑ πρέπει να λαμβάνει υπόψη του φυσικά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μέχρι τώρα δεν το κάναμε γιατί βασιζόμασταν σε ένα σχετικά παλαιό σύστημα, ίσως και πεπαλαιωμένο και πρέπει να πάρουμε υπόψη μας περισσότερες τεχνολογικές εξελίξεις. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι τόσο τεχνικό όσο πολιτικό και γι' αυτό πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση. Νομίζω όμως ότι πρέπει επίσης να μειωθούν τα διοικητικά κόστη και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν ένα απλοποιημένο σύστημα που να επιτρέπει διευκόλυνση του ενδοκινοτικού εμπορίου. Ευχαριστώ. Και η κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις ιδέες τους Τις περισσότερες, με τις περισσότερες συμφωνώ. Με, με άλλες όχι. Αλλά δέχομαι τις προτάσεις του κυρίου Κρόιτσμαν για την επίτευξη καλύτερου συντονισμού με τους κανόνες του κυρίου Ντεκάμπος για την τυποποίηση των τιμολογίων και γι' αυτό θα δεχτώ τις σχετικές τροπολογίες. Για τις απάτες συμφωνώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά εδώ είναι γνωμοδότηση και είμαι μέλος και της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολιτισμού και ξέρω ότι και εκείνοι γράφουν μια γνωμοδότηση σχετικά. Γι' αυτό δεν το even έφερα εγώ εδώ. Θα το πούν εκείνοι για τις απάτες. Εγώ μίλησα ε, με άποψη της εσωτερικής αγοράς. Στις 20 Ιουλίου λίγη διορία κατάθεση τροπολογιών. Περιμένω λοιπόν μέχρι τότε τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε 31 Αυγούστου. Και αυτό μου θυμίζει να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και πάλι τους διερμηνευτάς. Τους εύχομαι και αυτούς καλές διακοπές. Στις 31 Αυγούστου, Τρίτη στις 9 το πρωί θα ξαναβρεθούμε. Ελπίζω μέχρι τότε να έχετε αναπαυτικές διακοπές και μην ξεχάσετε να καταθέσετε τροπολογίες. Μέχρι τις 18, 19, 20 την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Γράψτε τις τροπολογίες και μετά να πάτε διακοπές. Ευχαριστώ και την κυρία Ράπτη γιατί ευχόμαστε ιδιαίτερα στους εισηγητές μας καλές διακοπές και καλύτερη εκδοχή των εκθέσεών τους όταν επιστρέψουν. Σας εύχομαι όλους καλησπέρα.